Dear colleagues, I think we, we will start hoping that the, the, the rest will join us. Ελπίζω λοιπόν ότι uh, οι υπόλοιποι θα έρθουν και ας ξεκινάμε θα έλεγα αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, είσαστε πάρα πολύ δυνατά και θα έλεγα να σταματήσετε να μιλάτε μεταξύ σας για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Και όποιος, ε, δεν θέλει, να, όποιος θέλει να μιλήσει κατηδία να ε, εγκαταλείψει την αίθουσα. Αρχικά έχουμε το ρόλο της πολιτικής συνοχής στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρώπη 2020 του Νούνο Τεξέρα και καταρχήν θα ήθελα να παρουσια... παρακαλέσω τον εισηγητή να παρουσιάσει την έκθεσή του και θέλω να σας πω ότι εδώ έχουμε δύο πολύ ενδιαφέροντες ομιλητές τον ε, Πέντρο Σόλβες Μύρα, ο οποίος, ε, εάν θυμάμαι καλά, δημιούργησε έναν νέο οργανισμό πολύ σημαντικό και έχουμε επίσης την έκθεση που μας ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Επιτροπός Μπανιά να καταρτήσουμε για την ενιαία αγορά και είναι εδώ η ε, Άννα Πάολα Λέισι του, η οποία είναι υπεύθυνη για το συντονισμό της πολιτικής των απομακρυσμένων πολιτικών για την Γενική Διεύθυνση ε, ε, Περιφερειών και δίνω το λόγο στον εισηγητή καταρχήν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να επισημάνω ένα ζήτημα που είναι αμυγός διαδικαστικό και αφορά κάτι άνευ στη δική μας επιτροπή, παρόλο που το είδαμε σε άλλες επιτροπές. Σήμερα θα έχουμε τη συζήτηση ενό εγγράφου εργασία Πορτογάλου συναδέλφου και θα ήθελα να εκφράσω την έντονή μου διαμαρτυρία γιατί δεν έχω διερμηνία από τα πορτογαλικά. Μου έχει ξανασυμβεί στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, για παράδειγμα. Και το επιχείρημα ήταν ότι δεν ήμουν τακτικό μέλο. Γι' αυτό δεν ήταν υποχρεωμένοι να μου εξασφαλίσουν ε, διερμηνία από τα πορτογαλικά. Στην Επιτροπή μας όμως ουδέποτε δεν συνάντησα τέτοιο φαινόμενο γιατί είμαι τακτικό μέλος και δεν φανταζόμουν ότι δεν θα υπήρχε διερμηνία για μένα. Υπάρχουν άνθρωποι που έκαναν 3.000 χιλιόμετρα για να έρθουν από τη Μαδέρα να παρακολουθήσουν τη συζήτηση και είναι πραγματικά παράδεκτο να έχουμε τόσες γλώσσες και να μην έχουμε πορτογαλικά για να ακούσουν αυτοί οι άνθρωποι τη μητρική του γλώσσα. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, αλλά ποια είναι τα κριτήρια επιλογής. Φαντάζομαι ότι κάποιος θα πρέπει να στερείται τη διερμηνία, αλλά με ποια λογική, με τι κριτήρια επιλογής ε, έχουν ορισμένη διερμηνία και άλλοι όχι. Θα ήθελα, εν πάση περιπτώσει, να ευχαριστήσω τη γραμματεία της Επιτροπής ε, που με βοήθησε, ε, ιδιαίτερα η Κάρλα Καρβάλιο, που από την αρχή με βοήθησε στην προετοιμασία της συζήτησης και της έκθεσης. Και θα ήθελα άλλη φορά να μην υπάρχουν τέτοια κενά. Εν πάση περιπτώσει, περνάμε στο κυρίω θέμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους, ε, τον, τον Πέδρο Σόλβεστη και την κυρία Άννα Πάουλα Λεσί. Τους ευχαριστώ θερμά που δέχτηκαν την πρόσκληση. Ε, για μένα είναι μεγάλη τιμή και προνόμιο η παρουσία τους εδώ Επίση, ε, θεωρώ τιμή μου και προνόμιο το γεγονό ότι έχουμε την ευκαιρία σήμερα στην Επιτροπή μας ε, να θέσουμε επιτάπητος ένα τόσο σημαντικό ζήτημα για μένα, που είναι το θέμα των εξόχως απόκεντρων περιοχών και το μέλλον της πολιτικής συνοχής στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το 2020. Θα ήθελα από την αρχή να επισημάνω ορισμένα σημεία τη ομάδα εργασία που θα αποτελέσουν, φαντάζομαι, και το αντικείμενο τη ανταλλαγή απόψεων. Οι εξόχω απόκεντρε περιοχέ, όπω ξέρετε, αυτή τη στιγμή είναι 9, θα γίνουν 8 εντός ολίγου από τον Ιανουάριο του 2012 και θα φέρει μία και είναι ε, περιοχές που έχουν ιδιαιτερότητες και που έχουν αναγνωριστεί στο άρθρο 349 της Συνθήκης. Το άρθρο 349 της Συνθήκης επιτρέπει διαφοροποιημένη μεταχείριση και την, ε, παρε... τις παρεκκλήσεις, τις εξαιρέσεις ε, από, πολλέ, πολλούς κοινοτικού κανόνες για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και περιλαμβάνονται εξαιρέσεις και σε σχέση με την πολιτική συνοχή. Στόχος μας είναι να υλοποιήσουμε τους στόχους της στρατηγικής του 2020 για αηφόρο ε, και ευφυή ανάπτυξη και στις εξόχως απόκεντρες περιοχέ. Θα ήθελα να συνοψίσω λίγο το έγγραφο εργασία μου σε τρει άξονε και προτεραιότητε. Η πρώτη είναι να προωθήσουμε διαφοροποιημένη και συνολική μεταχείριση των εξόχων και κοινή αντιμετώπιση των εξόχων απόκεντρων περιοχών, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητε των εξόχων απόκεντρων περιοχών στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, με ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτική τη συνοχή. Δεύτερη προτεραιότητα είναι η προσαρμοσμένη εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών ε, στις εξόχως απόκεντες περιοχές, πάλι προκειμένου να ληφθούν υπόψη ιδιαιτερότητες, αλλά και ο πλούτος που συνιστούν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τρίτη προτεραιότητα είναι να ε, βελτιωθεί η ενσωμάτωση των εξόχως απόκεντρων περιοχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις οικίες γεωγραφικές περιοχές, προωθώντας τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες και τις ε, χώρες που έχουν προνομιακούς δεσμούς ε, ιστορικούς και πολιτιστικούς. Στη συνθήκη της Λισαβόνας υπάρχει και μία ρήτρα πασαρέλα που επιτρέπει τη συμπερίληψη ή αποχώρηση ορισμένων περιοχών από το χαρακτηρισμό αυτό, όπως θα συμβεί με το Σάμπαρ Μπαρτελεμή. Άρα επιτρέπεται λοιπόν και η αποχώρηση ε, ορισμένων περιοχών από το χαρακτηρισμό των εξώχος απόκεντρων, αλλά και η συμπερίληψη. Αυτό είναι θετικό, γιατί μπορεί να επιτρέψει την είσοδο ε, υπερπόντιο διαπερισμάτων και άλλων χωρών μελών, του Σαρούμπας, για παράδειγμα, που είναι ολλανδική, ε, ολλανδικό διαμέρισμα και ε, μάλιστα θα διοργανωθεί εντό ολίγου δημοψήφισμα στην Αρούμπα. Οι πολίτε θα επιλέξουν αν θέλουν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο με τι εξόχω απόκεντρε περιοχέ τη Ευρώπη. Έτσι θα ενισχυθεί και το λόμπι των περιοχών αυτών εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη συμπερίληψη μια νέα περιοχή. Είναι η μοναδική ευκαιρία ε, τη συζήτηση αυτή και για άλλο λόγο, γιατί εξετάζουμε τι προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή ό,τι αφορά του κοινοτικού κανονισμού που θα διέπουν την πολιτική συνοχής και τα διορθωτικά ταμεία για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τα μέχρι στιγμής μηνύματα δεν είναι και πολύ θετικά. Για παράδειγμα, ε, το συγκεκριμένο δημοσιονο... Ε, ποσό του ΦΕΝΤΕΡ για τις εξόχους ε, απόκεντρες και τις αεροκατοικημένες περιοχές της Βόρειας Ευρώπης θα υποστεί μια μείωση. Αν συγκρίνουμε με το 2007-2013, την περίοδο 2014-2020, έχουμε μείωση κατά 976 από 976 σε 926 εκατομμύρια ευρώ. 50 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα λοιπόν, ε, δηλαδή 5% μείωση του προϋπολογισμού για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τις αεροκατοικημένες περιοχές. Σε ό,τι αφορά το στόχο ανταγωνιστικότητα και α, ε, επασχόληση, αν συγκρίνουμε με το προηγούμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, έχουμε 55 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου, ενώ για την επόμενη περίοδο είναι 53 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2014-2020, δηλαδή μείωση 3 περίπου το 100. Ε, είναι δύσκολο να εξηγήσουμε στους κατοίκους των εξόχως απόκεντρων περιοχών, που είναι από τους πιο φτωχούς της Ένωσης, ότι το ειδικό ποσό για αυτούς στο επόμενο πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο θα μειωθεί κατά 5%. Ενώ ε, για τις πιο πλούσιες και ευήμερες ε, περιοχές της Ένωσης, ε, που συγκεντρώνουν πάνω από 300% του μέσου όρου του ΑΕΠ, η μείωση είναι πολύ μικρότερη, είναι της τάξης του 3%. Πώς θα το εξηγήσουμε αυτό στους συμπολίτες μας. Είχαμε πολλές ανακοινώσεις, μελέτες, εκθέσεις τα τελευταία χρόνια που ασχολήθηκαν με το ζήτημα των από κέντρο περιοχών, αλλά η προσέγγιση γίνεται κυρίως θεωρητικά και το ποιοτικό άλμα που σήμανε για την Ευρωπαϊκή Ένωση η έκθεση Solves ε, συνίσταται ότι για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ένα έγγραφο που μας δείχνει την κατεύθυνση τη σωστή άγουσα, έναν οδικό χάρτη που επισημαίνει τα προβλήματα, τις αδυναμίες ε, των εξόχων απόκεντρο περιοχών, αλλά περιλαμβάνει και συστάσεις, 22 συστάσεις αν δεν κάνω λάθος, με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για το μέλλον. Σε ό,τι αφορά αυτή την έκθεση, σημαντικό ε, ζητήμα ε, αποτελεί η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις ε, περιοχές αυτές. Ο Φεντέρ, το ΦΕΝΤΕΡ προβλέπει για τέτοια περίπτωση στη χρηματοδότηση 50%. Ο Επίτροπο Ιωάννης Αν πρόσφατα στη Μαρτινίκα, στη, στο συνέδριο των εξόχων απόκεντρων περιοχών, είπαν ότι όσοι θέλουν να κρατήσουν το ειδικό, το ειδικό ποσό του προπολογισμού θα έπρεπε να δώσουν μεγάλη μάχη, μακροχρόνια μάχη στο Συμβούλιο. Αυτά ήταν τα λόγια του Επιτρόπου. Δεν ξέρω ποια θα είναι η μάχη στο Συμβούλιο. Πάντως, ε, εγώ είμαι έτοιμος να ξεκινήσω εδώ τον πόλεμο, εντός της Επιτροπής ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ δεν θέλω απλώ να διατηρηθεί αυτό το κονδύλιο, αλλά θέλω να αυξηθεί κιόλα. ε, ένα επιχείρημα ε, που αναφέρεται είναι η χαμηλή απορρόφηση των ε, κονδυλίων αυτών. Με τη συγχρηματοδότηση όμως 50% που προβλέπεται από το ΦΕΝΤΕΡ, πώ ε, θα ανταπεξέλθουν στι υποχρεώσει του στα κράτη-μέλη που ήδη αντιμετωπίζουν κρίση, πολλό δε μάλλον οι εξόχω απόκεντρε περιοχέ που είναι σε ακόμη δυσμενέστερη κατάσταση. Ε, με βάση τις συστάσεις του κυρίου Σόλβες, εγώ θα πρότεινα το ποσοστό χρηματοδότησης από αυτό το συγκεκριμένο ποσό να περάσει από το 50% σε 85%, όπως ισχύει για άλλες περιπτώσεις του ΦΕΝΤΕΡ. <clears throat> Νομίζω ότι έτσι θα βοηθούν οι περιοχές αυτές να απορροφήσουν καλύτερα τα κονδύλια. Κάτι άλλο ε, που θα πρέπει να θέσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη Γενική Διεύθυνση Ρέτζι, είναι αυτό, γιατί οι εξόχως απόκειτες ε, περιοχές θα πρέπει να τύχουν τις ε, προσοχή που αξίζουν και θα πρέπει να δώσουμε, να διεκδικήσουμε έναν ε, ηγετικό ρόλο. Και νομίζω ότι η Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο θα πρέπει αυτή να αναλάβει αυτή την ευθύνη και τον ηγετικό ρόλο. Αυτό θα κρίνει το κατά πόσο θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε εμπράκτος αυτές τις 22 συστάσεις που περιλαμβάνει η μελέτη του κυρίου Σόλβες. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή την ε, πρωτοβουλία από την Γενική ε, διεύθυνση Ρέτζιο και δεν θα μακρηγορήσω άλλο, προτιμώ να ακούσουμε τους προσκεκλημένους εμπειρογνώμονε μας για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Thank you ε, very much indeed. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, καλό τον Πέτρο όλες να μας μιλήσει πάνω στα κυριότερα κατά τη γνώμη του σημεία της έκθεσης σχετικά με την πολιτική για να καταλάβουμε καλύτερα περί τίνος πρόκειται. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα επιχειρήσω σε σύντομο χρονικό διάστημα να σας παρουσιάσω τα θεμελιώδη στοιχεία της έκθεσης. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω και την Πρόεδρο της Επιτροπής και τον ε, εισηγητή για την πρόσκλησή τους. Όπως ξέρετε, στις 12 Οκτωβρίου επέδωσα την έκθεση στους επιτρόπου Μπαρνία και Χάν και είναι πλέον ε, πρόσθετη και μπορείτε να τη διαβάσετε. Θα ήθελα να επισημάνω ορισμένα θεμελιώδη στοιχεία της έκθεσης. Όλη η προσπάθεια και όλο το έργο ε, ήταν μια ανάθεση του Επιτρόπου Μπαρνιέ προκειμένου να εξεταστεί ο αντίκτυπος εσωτερικής αγοράς και η αποτελεσματικότητά της στις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Εγώ διορίστηκα το Μάιο και εργάστηκα μέχρι το Σεπτέμβριο εκπονώντας την έκθεση. Το πρώτο που ε, μας προβλημάτισε στην έκθεση είναι η διαφοροποίηση μεταξύ της θεωρίας της ενιαίας αγοράς και της πραγματικότητας έμπρακτης εφαρμογής της ενιαίας αγοράς στις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Γιατί ε, το να πιστεύουμε ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε την ενιαία αγορά όπως την σχεδιάσαμε σε περιορισμένες σε μικρές περιοχές ή σε εξόχως απόκεντρες περιοχές που δεν έχουν μεγάλη διασύνδεση με υπόλοιπε περιοχές της υπηρετικής Ευρώπης είναι εσφαλμένο. Δείχνει άγνοια για τα πραγματικά προβλήματα των εξόχως απόκεντρων περιοχών. Νομίζω ότι ήταν σκόπιμη και κατάλληλη αυτή η έκθεση καθώς και εύστοχη γιατί υπήρχε ζήτηση, έπρεπε να δούμε τι θα κάνουμε. Ο Μάριο Μόντις όταν το Μάιο υπέβαλε την, το 2010 την πρόταση για την εσωτερική αγορά είπε ότι είναι λιγότερο δημοφιλής από ποτέ η πρόταση αλλά περισσότερο κατάλληλη και σκόπιμη από ποτέ. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση αυτή. Στην ανάλυση και τη διάγνωση των προβλημάτων για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές ε, το θέμα δεν είναι να κρατήσουμε την παρελθούσα κατάσταση και να κάνουμε έναν κατάλογο παραπώνων. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κάνουμε μια κριτική ανάλυση και να διαπιστώσουμε ποια στοιχεία της εσωτερικής αγοράς και της νέας οικονομικής πραγματικότητας μπορούν να μας βοηθήσουν να ανοίξουμε νέους δρόμους. Θα ήθελα να επισημάνω κάποια αναφυσβήτητα στοιχεία. Καταρχήν, η πραγματικότητα, η καθημερινότητα των εξόχων από, από, από μακροπεριχών η απομάκρυνσή τους, η απόσταση, η μεγάλη απόσταση, οι καιρικέ ε, συνθήκες, η μορφολογία. Όλα αυτά είναι διαφορετικά. Σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, εκεί υπάρχουν κάποιες καινοτομίες. Αναφυσβήτητα το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η ίδια η κρίση. Η κρίση αυτή είχε τεράστιο και πολύ αρνητικό αντίκτυπο στις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Ιδιαίτερα έπληξε την απασχόληση, το επίπεδο απασχόληση. Αλλά δημιουργήθηκαν και νέα ευκαιρίε, ιδιαίτερα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική και το 2020. Εκεί ε, στοιχεία όπω η αηφόρος ανάπτυξη, η μεγαλύτερη προσοχή του για το περιβάλλον, ε, καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι πολύ σημαντικά και για τις ε, εξόχως απόκεντρες περιοχές. Είπα λοιπόν ότι είναι και σκόπιμη και κατάλληλη αυτή η στιγμή για την υποβολή της έκθεσης, γιατί όπως είπε και ο κύριος Τεσέρα, αυτό που ε, ζούμε σήμερα είναι μια συζήτηση για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Και εκεί προσπαθούμε με αποτελεσματικό τρόπο να προσαρμόσουμε τους πόρους στις, ε, στους, στους στόχους μας. Και αυτό θα ισχύσει και για τις εξόχως απόκειτες περιοχές. Εγώ δεν θα επισέλθω στη συζήτηση, στην ουσία της συζήτησης για τους πόρους, ούτε θα σχολιάσω τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό. Τέτοια σχόλια δεν έχουν τη θέση τους εδώ. Με την έκθεσή μου, εγώ ήθελα να προτείνω κάποιες νέες ερμηνείες και να περάσουμε σε διαφορετική αντίληψη για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Αντί να τις βλέπουμε ε, με τα στοιχεία του παρελθόντος ε, και με ένα στιγμιότυπο που στόχο έχει να διατηρήσει την προηγούμενη κατάσταση, προτείνω μία ε, ανατένιση του μέλλοντος. 22 είναι οι συστάσεις που κατέθεσα, που περιορίζονται σε 7 άξονες και στόχος αυτών των 22 συστάσεων είναι να εντοπίσουν κάποιο καινοτόμα σημεία και νέες προκλήσεις για τις υπεραπόκεντρες περιοχές που μπορεί να ενδιαφέρουν για το μέλλον. Το πρώτο ζήτημα είναι φυσικά το θέμα της χρηματοδότησης. Της χρηματοδότησης γενικά, αλλά της χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ειδικότερα. Πρόκειται για κατακαιρματισμένες αγορές. Και μέχρι με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς από τις μεγάλες πόλεις, με τα προβλήματα που δημιουργούνται. Και παρόλο που επίσημα η ελευθερία διακίνησης των πολιτών υπάρχει στα χαρτιά, η κινητικότητα των πολιτών των εξόχως απόκεντρων περιοχών είναι σχετικά περιορισμένη. Και είναι αλήθεια ότι σε ορισμένες περιπτώσεις κάποια στοιχεία δεν ευνοούν την αύξηση της κινητικότητας αρκεί να δούμε τι προγράμματα εφαρμόζουμε για την κινητικότητα νέων και φοιτητών και πώς προσαρμόζονται στις ανα... ανάγκες αυτών των περιοχών. Δυστυχώ δεν ανταποκρίνονται ούτε η κατάρτιση, τα προγράμματα κατάρτιση ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις των νέων τεχνολογικών. Και υπάρχει και ένα εξάρτηση των περιοχών από το ευρύτερο περιφερειακό πλαίσιο. Τρίτος άξονας, ανάγκη βελτίωσης της εμπιστοσύνης του καταναλώτη και ιδιαίτερα του εργοδότη, προκειμένου να διαθετηθούν οι διαφορές μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των κοντινών περιοχών. Υπάρχουν τέτοιε ορισμένες φιλονικίες, άλλες φορές είναι πραγματικές φιλονικίες, άλλες φορές είναι έλλειψη διαδικασίας για αποτελεσματικότερη συνεργασία. Άλλο σημαντικό σημείο είναι ανάγκη ε, εφοδιασμού των περιοχών αυτών με τις απαραίτητες υποδομές και για την πρόσβαση στο, σε, στην κοινοτική και εξωκοινοτική επικράτεια, αλλά κυρίως ε, για να προσαρμοστούν στις προκλήσεις ε, των νέων τεχνολογιών. Θέλουμε φυσικά <coughs> δίκτυα συγκοινωνιών, αλλά κυρίως προσπελασιμότητα, ε, η πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες. Κάτι που σημαίνει ειδικά δίκτυα για να ε, βελτιωθεί αυτή η πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες. Πέμπτος άξορας είναι η συμπερίληψη της Ρού στην ενιαία ψηφιακή αγορά. Ένα σημαντικό στοιχείο της RUT μέχρι στιγμής ήταν η γεωγραφική κατάσταση αυτών των εξόχως απόκεντρων περιοχών που δεν τους επέτρεπαν να ενταχθούν σε ε, δραστηριότητες της υπηρετικής Ευρώπης. Στον ψηφιακό κόσμο όμως ε, το θέμα της ε, απόστασης δεν ε, μετράει αρκεί να υπάρχουν τα κατάλληλα δίκτυα που να επιτρέπουν την επικοινωνία. Δηλαδή, στο μέλλον η αγορά που θα στηρίζεται όχι τόσο στα εργατικά χέρια, αλλά στις δεξιότητες ε, και θα εξυπηρετήσει υπηρεσίες, θα είναι η αγορά του μέλλοντος. Θα δούμε λοιπόν από πού θα περνάνε οι μεγάλοι διάβλοι επικοινωνία και το ε, θέμα της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών θα ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις εξόχως κεντρές περιοχές. Ένα άλλο θέμα αφορά την καλύτερη χρήση των ενεργειακών πόρων. Το πρόγραμμα για το 2020, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική, αναφέρεται ως κεφαλαιόδου σημασία η χρήση των ανανεώσιμων ποιών ενέργειας και άρα η μείωση των, της εκπομπής καυσαερίων. Τα νησιά σίγουρα από αυτήν την άποψη μας προσφέρουν πολλές α, δυνατότητες. Καταρχήν ενδιαφέρονται και τα νησιά για τη μείωση των εκπομπών αεριοθερμοκηπίου, αλλά και σε πολλά νησιά έχουμε πολλά στοιχεία ε, που θα μας επιτρέψουν να σημειώσουμε πρόοδο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για παράδειγμα, έχουμε το πιλωτικό πρόγραμμα του, της νήσους Γέρο, αλλά και από την ανταλλαγή εμπειριών που είχαμε από προγράμματα όπως το Σύμφωνο των Νήσων, θα μας επιτρέψουν να δούμε πώς ε, θα κατορθώσουμε να μειώσουμε κατά 20% τα επίπεδα των καψαρίων ε, σε σχέση με το 1990. Πιστεύω ότι τα νησιά θα καταφέρουν να υλοποιήσουν αυτό το στόχο για το 2020 και μάλιστα και με ανταγωνιστικό τρόπο. Η μείωση από την ενεργειακή εξάρτηση είναι ένα από τα στοιχεία που επίσης θα τύχουν προσοχής. Άλλο στοιχείο που επίσης ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και είναι ο έβδομος άξονας αφορά την κοινωνική συνοχή. Μέσω της ε, ε, εμπέδωσης και βελτίωση των, μέτρων, των ειδικών μέτρων για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές προκειμένου να έρθουν τα εμπόδια στη συμμετοχή στην, τη συμμετοχή στην ενιαία αγορά. Πολιτική συνοχής, ε, ΠΟΣΕΗ γεωργικό, για τα γεωργικά προϊόντα και ούτω καθεξής. Σίγουρα υπάρχουν πολλές ε, ιδιαιτερότητες και θα πρέπει να αξιοποιηθούν. Τώρα, τι θα πρέπει να γίνει σε περίπτωση βιοπικιλότητας ε, ή καταπολέμησης ε, κλιματικών αλλαγών. Και τα θέματα αυτά είναι σημαντικά για τις εξόχως απόκεντρε περιοχές, ιδιαίτερα αν τα δούμε υπό το πρίσμα της καινοτομία και των επενδύσεων και τις σπουδαιότητες που έχει η θάλασσα για τις ε, υπεραπόκεντρες περιοχές. Εκτός από τους επτά άξονες, να προσθέσω και δύο σχόλια και να ολοκληρώσω. Θέλουμε να αναβαθμίσουμε το ρόλο ή την εξωτερική διάσταση της ενιαίας αγοράς, και επίσης ε, ανάγκη να εξετάσουμε περιφερειακά προγράμματα γειτονίας. Πολλές φορές οι υπεραπόκεντρες αυτές ε, περιοχές ξεχνούν ε, το φυσικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. Εστιάζονται κυρίως στις σχέσεις με την περιοτική Ευρώπη. Είναι σημαντικά λοιπόν και τα περιφερειακά προγράμματα, σχέδια γειτονίας. Γιατί μερικές φορές η αντίληψη που έχουμε για τη συνεργασία με τα άλλα εδάφη, διαμερίσματα και εξόχως απόκεντρε περιοχές είναι σημαντική γιατί και εκεί υπάρχει χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης και μερικές φορές παρόλο που υπάρχει δυνατότητα και διαθέσιμα κονδύλια δεν εφαρμόζονται εξαιτία της έλλειψης συντονισμού ε, διαπεριφερειακά μεταξύ αυτών των περιοχών. Επαναλαμβάνω δύο ακόμη σχόλια. Οι εξόχως απόκεντρε περιοχές θα πρέπει να γίνουν οι πύλε τη Ευρώπη η πύλη της Ευρώπης προς την Αμερική και προς την Αφρική, νοτίως και δυτικά, και επίσης να δώσουμε έμφαση σε κάποια εγκάρσια μέτρα, να συμπεριλάβουμε ε, ανάλυση του αντικτύπου και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές για οποιαδήποτε μέτρα, οποιαδήποτε μέτρα εξετάζουμε και να καταστήσουμε πιο ορατές αυτές τις περιοχές και να τις λάβουμε υπόψη στις διάφορες δράσεις στρατηγικής του 2020. Η ενιαία αγορά λοιπόν για βελτίωση, ως μηχανισμός για τη βελτίωση των ανταλλαγών για την υλοποίηση της υφόρου ανάπτυξης και της αναβάθμισης του βιωτικού επίπεδου των Ευρωπαίων πολιτών ε, είναι σημαντική και το δυναμικό της θα φανεί ιδιαίτερα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές όπου προς το παρόν μένει σχετικά αναξιοποιητό. Θα δούμε τώρα τι προβλήματα υπάρχουν και τι ε, λύσεις θα προταθούν. Στόχος εκθεσής μου είναι να στραφεί προς το μέλλον και άσχετα με το, δημοσιονομικό σκέλος αναζητούμε κάποιες καινοτόμες λύσεις για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές για να αξιοποιήσουμε το δυναμικό τους και τις νέες τους δυνατότητες και μετά φυσικά θα εξαρτηθεί από την Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πώς θα συνεχίσουν αυτό το έργο και κυρίως πώς θα συμφιλιώσουν το στόχο ανάπτυξης των περιοχών αυτών με το νομικό πλαίσιο και την σχετικά μικρή ε, διαθεσιμότητα των δημοσιονομικών πόρων. Ευχαριστώ. Thank you. We Ευχαριστώ. Θα ακούσουμε την ε, Πάολα Λέση πρώτα και μετά θα γίνει συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Με συγχωρείτε, θα μπορούσα να μιλήσω και πορτογαλικά, αλλά νομίζω ότι θα είμαι πιο άνετη να μιλήσω γαλλικά και γι' αυτό θέλω να ζητήσω συγγνώμη από αυτούς που ήρθαν από την Πορτογαλία και δεν έχουν μετάφραση προς τη γλώσσα τους. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι ε, όσον αφορά τις ακραίες περιφερικές περιοχές εσείς φροντίσατε να μπορέσει να υπάρξει μία επέμβαση και η Επιτροπή οθέτησε ε, δύο <clears throat> ανακοινώσεις σχετικά με αυτή την περιοχή και γι' αυτό θέλω να χαιρετήσω αυτή την κίνησή σας. Θέλω επίσης να χαιρετήσω τον Ευρωβουλευτή κύριο Τεσέρα, ο οποίος μας είπε ε, τι είναι τα προβλήματα και τι θα γίνει με το φιλοπορίας το οποίο παρουσιάζει όλα τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και όλες τις πτυχές που θα πρέπει να επιληθούν και να ρυθμιστούν τους επόμενους μήνες. Καταρχήν θα ήθελα να παρουσιάσω τη μονάδα μου. Είμαστε μία μικρή ομάδα στην Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο που συντονίζει τις κοινοτικές πολιτικές για τις διάφορες εξόχως απόκεντρες περιοχές και ε, όπως είπε και ο κύριος Τεσέρα το θέμα το δημοσιονομικό μας διαφεύγει δηλαδή δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε προτάσεις σχετικά με το πολιετές δημοσιονομικό πρόγραμμα για το μέλλον και γι' αυτό λυπούμαστε ιδιαίτερα ότι οι πολιτικές αυτές, εγώ τουλάχιστον λυπούμε πολύ γιατί οι προτάσεις οι οποίες αναφέρονται σε αυτές τις εξόχως απόκεντρες περιοχές ε, σημείωσαν μία μείωση χρηματοδότησης. Αλλά Πρέπει να σας πω ότι η μείωση αυτή αντικατοπτρίζει τις δημοσιονομικές περικοπές τις οποίες επέβαλαν οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη και να διατυπώσει μία πρόταση στα πλαίσια της, των δημοσιονομικών προοπτικών σε χαμηλότερο επίπεδο από ό,τι στο παρελθόν αλλά και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ βασικό και πρέπει να σημειωθεί. Το είπατε άλλωστε ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αυτό το οποίο λέει και οι λέξεις, δηλαδή προτάσεις. Τώρα πρέπει να γίνει πάρα πολύ εργασία και με το Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο κατά τρόπον ώστε οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις οι οποίες θεωρούνται σημαντικές να μπορέσουν να γίνουν διότι κατά το 2012-2013 κατόπιν ε, των διαπραγματεύσεων θα μπορέσουν να καταρτιστούν προτεραιότητες για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις οι οποίες προκύπτουν. Ξέρω βέβαια ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος και η συζήτηση θα μπορούσε να είναι πολύ πιο εμπεριστατωμένη από τα λίγα που θα πω εγώ εδώ αλλά θέλω να τονίσω ότι η πολιτική συνοχής και τις προτάσεις που έγιναν προενός μηνός ε, διότι βρίσκονται στο επίκεντρο της ε, ευρωπαϊκής στρατηγικής και η πολιτική ε, συνοχή είναι ένα από τα μέσα βάσει των οποίων προσπαθούμε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, να διατυπώσουμε συγκεκριμένα μέτρα για τη βιώσιμη έξυπνη ανάπτυξη που απευθύνεται σε όλους και αυτό πρέπει να σημειώσουμε για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, πέραν των δημοσιονομικών στόχων. Ε, νομίζω ότι οι περιοχές αυτές το γνωρίζουν και έχουν σημειώσει αυτή τη μείωση ε, του του προπολογισμού και ο Επίτροπος Γιωχάνες Χάν στην ε, συνεδρίαση η οποία έγινε ε, ε, άκουσε τις απόψεις όλων των εκπροσώπων των αποκέντρων περιοχών στη συνέντευξη της Μαρτινίκας και σημείωσε όλες τις αντιδράσεις της προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμφωνώ δε με το ότι πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Ε, Λέχει αυτό στην ανακοίνωση, έχουμε αναφερθεί σε ορισμένες δράσεις και ε, εγώ τουλάχιστον προσπάθησα να είμαι πιο συγκεκριμένος και να υπάρξουν ορισμένες ε, ανακοινώσεις ε, οι οποίες καταρτίζονται για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στην ανακοίνωση αυτή θα ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν ε, είτε είναι στρατηγικά είτε είναι πολιτικά. Εγώ βέβαια θα ξεκινήσω από την έκθεση Σολβές η οποία είναι πολύ σημαντική και την οποία μελετούμε και εξετάζουμε για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να την υλοποιήσουμε μέσω της ανακοίνωσής μας. Υπάρχει όμως και το έγγραφο το οποίο έχει καταρτιστεί ε, για τους ευρωβουλευτές μέλη των ε, εξόχως από κέντρων περιοχών και ε, θα πρέπει να συνεννοηθείτε και με τον υπεύθυνο επίπεδο, ε, επίτροπο Χάν για να μπορέσετε ε, να προβάλλετε τις θέσεις σας. Το έγγραφό μας νομίζω ανταποκρίνεται εις τις ανάγκες και στις προσμονές των εξόχως από κέντρων περιοχών και είναι το αποτέλεσμα μιας εργασίας στην οποία κατήρτισε η μονάδα μου σχετικά με την ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Και ε, βάσει της εκθέσεως του Υπουργού Πέντρο Αλβες ο οποίος γνωρίζει ότι έχει καταρτιστεί το έγγραφο αυτό, όλα αυτά μαζί αποτελούν ένα σύνολο που τονίζει τη σημασία των εξόχως αποκέντρων περιοχών κατά τρόπον ώστε να διατυπωθούν προτάσεις οι οποίες να συνάδουν με τις προσδοκίες των περιοχών αυτών και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο σύνολό της. Δεν ξέρω πόσο χρόνο ακόμη <clears throat> έχω στη διάθεσή μου, θα ήθελα όμως να σας πω και θα το δούμε σχετικά με ε, τις ε, άλλες ε, τα άλλα θέματα ότι για μας είναι σημαντικό να παρακολουθούμε τις ε, εξόχως απόκεντρες περιοχές και προβλέπεται τη συνθήκη η αλλαγή καθεστώτος για ορισμένες περιοχές ήδη δε για τη μία έχει γίνει αυτή η αίτηση για τη Μαγιότ που είναι ε, ε, μια γαλλική περιοχή ε, εξόχως απόκεντρη και τώρα πρέπει να γίνει η εξέταση των στοιχείων από τη Γενική Διεύθυνση για να περιληφθεί αλλά υπάρχουν και άλλες περιοχές όπως η Αρούμπα και άλλες τις οποίες προαναφέρατε μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τίποτα το επίσημο αλλά μόλις θα υποβληθούν επισήμως οι αιτήσει θα τα εξετάσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Ε, επίσης πιστεύω ότι ό,τι ήταν ουσιαστικό ελέγχθη από τον Πέντρο Σόλβες και το έγγραφο της, ε, ε της Επιτροπής του κυρίου Νούνο 4 αλλά ίσως αυτό που πρέπει να πω είναι ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις που απορρέουν από τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρώ ότι για το άμεσο μέλλον πρέπει να ενημερώσουμε τις απόκεντρες αυτές περιοχές να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην επόμενη φάση, δηλαδή να εμπλακούν στη λήψη αποφάσεων, να τους λεχθεί ότι πρέπει να δραστηριοποιηθούν στις ε, συμβάσεις συνεργασίες που θα διατυπωθούν στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής να δημιουργήσουν αυτή την διοικητική, τοπική, αυτό το δυναμικό το οποίο δεν υφίσταται ακόμη και να τονίσουμε ότι είναι πολύ σημαντικό για να υπάρξει κάθε δυνατή ανάπτυξη να υπάρχει το, το πρότυπο αυτό του έλικα, δηλαδή συμπληρωματικότητος, να υπάρχουν οι ομόλογοι από ε, τις πλευράς του δημοσίου, οι επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια ανάπτυξης, ο ακαδημαϊκός κόσμος, ο πανεπιστημιακός, η έρευνα, όλοι δηλαδή οι τομείς να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια. Και στα πλαίσια αυτά θα ήθελα εδώ να ακολουθήσω αυτά που είπε ο Πέντρο Σόλβες ε, σχετικά με την καινοτομία, με το πώς μπορούμε να το του ό,τι ήδη υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκφράσει τη συμφωνία της για να ε, καταρτήσει τους στόχους της και να δημιουργήσει ένα νέο στόχο, μία ειδική πλατφόρμα που θα απευθύνεται σε εξόχως απόκεντρες περιοχές για να μπορούμε να ξεκινήσουμε αυτή την εργασία και για τις περιοχές αυτές που έχουν κοινά προβλήματα και πολλές φορές επιζητούν κοινέ λύσεις να μπορέσουν ήδη να συμμετάσχουν στα ήδη υπάρχοντα και να μπορέσουν να προβάλλουν τις κινήσεις τους και τα επιτεύγματά τους. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι είναι σημαντικό για τις περιοχές αυτές να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μέτρο, το, το μέλλον και να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που είναι στη διάθεσή τους ε, διότι υπάρχουν τομείς ε, με, με πολύ υψηλή χρηματοδότηση αλλά και άλλοι τομείς ε, όπου διατίθεται χρηματοδότηση για την αναπτυξιακή έρευνα, για το ΣΥΠ που είναι το πρόγραμμα της καινοτομίας στις ανταλλαγές εκπαιδευτικών των φοιτητών ή άλλοι ακόμη τομείς όπου έχουμε ευελιξία για αυτή την περίοδο. Και τέλος θα ήθελα να σας πω ολοκληρώνοντας ότι θέλω να σας υπενθυμίσω ε, ενδέχεται να σας λέω κάτι το προφανές αλλά Ίσως ε, πρέπει να επωφεληθούμε τις ευκαιρίες που μας δίνεται τώρα, διότι βρισκόμαστε σε μία κρίσιμη περίοδο όπου θα μπορέσουμε να προβούμε στις αναγκαίες τροπολογίες και αλλαγές που οι απόμακρες περιοχές θεωρούν ως προτεραιότητες οι οποίες κάπως είχαν παραβλεφθεί. Δεν θα σας μιλήσω για τις επιτυχίες, έχουμε πολλές προτάσεις οι οποίες είναι πολύ θετικές και ίσως στα πλαίσια της συζητήσεως θα επανέλθω στις προτάσεις αυτές οι οποίες επέτρεψαν να ανταποκριθούμε σε ορισμένες δυσκολίες και ε, να επιλύσουμε διάφορα προβλήματα. Εάν λοιπόν θέλει η πρόεδρος ε, ε, θα, συμπληρώσω κατά τη συζήτηση. Ευχαριστώ Ανά Πόλα. Πέραμε σε ερωτήσεις, σχόλια. Να πω όμως προηγουμένως ότι έχει η σημασία να σκεφτούμε πώς όλα αυτά συνδέονται με το μελλοντικό νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τις ε, εξόχως απόκεντρες περιοχές. Να δούμε δηλαδή πώς αυτό το νομοθετικό κανονιστικό πλαίσιο θα μπορέσει να καταστήσει και τις πολιτικές αποτελεσματικές, όπως είπε και ο Φέντρο Σόλπες. Τέλος, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι πολύ ευγνώμων που συζητάμε το θέμα αυτό και ιδίω ε, είμαι πολύ ευγνώμων για τα σχόλια του κυρίου Σόλβες, ε, της κυρίας Λεσί και του, την εισήγηση του κυρίου Τεχέρα. Καταρχήν πρέπει να δούμε τι ε, ε, υπάρχει, ε, τι γνώση έχουμε και πώς πρέπει να ενισχύσουμε τις εξόχως απόκεντρες περιοχές στην Ευρώπη. Είχα συμμετάσχει εις την αποστολή στην Γαλλική και ε, πρέπει να διαπιστώσουμε ότι ε, υπάρχουν πολλές ελλείψεις εκεί και πρέπει να δούμε ε, πώς θα τις καλύψουμε. Επειδή όμως τώρα γνωρίζω αυτή την περιοχή, όπως άλλωστε και το νησί της Τενερίφης, γνωρίζω ότι αυτές οι περιφερειακές περιοχές δεν πρέπει να αξιολογηθούν βάσει των αδυναμιών τους, δηλαδή απόμακρες, απομονωμένες, δύσκολες μεταφορές, αλλά πρέπει να τονίσουμε και τα ισχυρά του σημεία, δηλαδή ε, τι προστιθέμενη αξία έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω αυτών των απομάκρων περιοχών ε, σε κλιματολογικές ζώνες οι οποίες είναι διαφορετικές από την Ευρωπαϊκή, οι οποίες μπορούν να ανταποκριθούν σε προκλήσεις ε, οι οποίες διαγράφονται σε άλλα μέρη του κόσμου και μπορούν έτσι να κοινοποιηθούν τα στοιχεία αυτά στην Ευρώπη κατά τρόπον ώστε με τις δυνατότητές μας να μπορέσουμε να τα επιλύσουμε και καινότομα να παρέμβουμε στην κλιματολογική προστασία, στην ενεργειακή ασφάλεια και σε άλλους τομείς για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις δυνατότητές μας. Ο κύριος Σόλβες άλλωστε αναφέρθηκε εις την εξάρτηση από καύσιμα στις περιοχές αυτές, ιδίω στην Τενερίφη, υπάρχει ένα Ινστιτούτο για ανανεώσιμες πηγές ενεργείας εδώ και χρόνια και το ερώτημα τίθεται πώς μπορεί κανείς ε, να χρησιμοποιήσει και να αξιοποιήσει τις ανανόσιμες πηγές ενεργείας ε, σε περιοχές υποτροπικές και τροπικές. Και αυτό αναφέρεται στις ανανεώσιμες πηγές ενεργείας. Το ίδιο είδα και στη Γαλλική ε, Ουγιάννα, γιατί είδαμε ότι υπάρχει πρόοδος, υπάρχει γυτνία με ε, τη ε, Βραζιλία και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Μητρόπολη, δηλαδή η Γαλλία σε αυτή την περιφερειακή της περιοχή. Ε, διότι ένα μέρος είναι στο υποτροπικό δάσος και ε, ε, υπάρχουν σημαντικότατες βροχοπτώσεις αλλά έτσι μπορούμε να προβούμε σε σημαντικές ε, έρευνες οι οποίες να χρησιμοποιηθούν και αλλού. Άρα αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν όσον αφορά την πολιτική προωθήσεως της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δηλαδή να προβαίνουμε σε κοινέ διαπιστώσεις με τους επιτόπου παράγοντες και να μπορούμε να τα αξιοποιούμε. Χωρίς να με παρανοήσετε, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές έχουν σαν άμεσο δαιμόνα την μητέρα χώρα τους. Αλλά εδώ έχουν διαγραφεί διάφορες δυνατότητες όπου σαν Ευρωπαίοι μπορούμε να παριστάμεθα μακρά της γεωγραφικής μας μας επικράτειας και ε, να στηρίξουμε προσπάθειες οι οποίες γίνονται και σε άλλα μέρη του κόσμου. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σάλβες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Νούνο Τεσέιρα, τον Επίτροπο Πέτρο Σόλβης και την κυρία Ναπαόλα Λάση για την παρουσία τους στην Επιτροπή μας και τη δυνατότητα που έχουμε για την ε, συζήτηση αυτή. Ο Επίτροπος Πέδρος Σόλβες ε, μας παρουσίασε μια έκθεση πολύ σαφή, αντικειμενική, με εστί και με πολύ συγκεκριμένες και σημαντικές προτάσεις για το μέλλον ε, της στρατηγικής για τις εξόχως από κέντρες περιοχές. Ίσως παρά είναι απτές και συγκεκριμένες αυτές οι προτάσεις για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που προτιμά πιο ενιολογικές και αφηρημένες εργασίες για τις εξόχως απόκεντες περιοχές προκειμένου να εξασφαλίσει μεγαλύτερο περιθώριο λιγμών. Πάντως πιστεύω ότι αυτή η έκθεση αποτελέσει σημαντικό εργαλείο εργασίας όταν θα εξετάσουμε την στρατηγική για τις εξόχως απόκεντες περιοχές. Θα ήθελα επίσης ε, να πω ότι στα πλαίσια του πακέτου που υποβλήθηκε ε, ήταν σημαντικό το σκέλος ε, των από απόκεντρων περιοχών και της αυτόνομης ε, πολιτικής συνοχής προκειμένου να εξελιχθούν οι μεγάλες ανισότητες μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών. Αυτό ευνοεί τις εξόχως απόκεντρες περιοχές για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους και να συγκλίνουν όλο και περισσότερο με την υπόλοιπη, με την υπηρετική Ευρώπη. Δεν μπορούμε να κλείνουμε την πόρτα ε, στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και να ανοίγουμε μια άλλη πόρτα με ρηξικέλευτες μεταρρυθμίσεις. Νομίζω ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε την προεργασία που έγινε και από αυτή την άποψη θα χρησιμοποιήσουμε ιδιαίτερα την πολιτική συνοχή. Η κυρία Άννα Παύλα Λάση είπε ότι όλοι οι πρόεδροι των υπεραπόμακρων περιοχών μίλησαν για την ε, η ε, ιδιαίτερη ε, σημασία που έχει το ΦΕΝΤΕΡ για να αντιμετωπιστεί το επιπλέον κόστος για τις ε, περιοχές αυτές. Νομίζω ότι όλοι θα επισημάνω αυτή την αρνητική πτυχή και για δύο πολύ απλούς λόγους. Καταρχήν, για να ε, αποκατασταθεί μία δικαιοσύνη θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τους χαρακτήρες ε, και η ευπάθεια αυτών των περιοχών. Δεν μπορούμε λοιπόν να περικόπτουμε περισσότερο τα κονδύλια για τις ε, ε, εξόχως απόκεντρες περιοχές, ενώ οι μειώσεις για άλλα ταμεία, για άλλες περιφέρειες είναι λιγότερο δραστικές. Δεν έχει νόημα κάτι τέτοιο. Είναι πολύ άδικο για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Κάτι άλλο που θα ήθελα να προσθέσω είναι το εξή. Υπάρχει προσανατολισμός και μία τάση για στόχευση των πολιτικών σε συγκεκριμένους στόχους προκειμένου να καταμετρηθεί η αποτελεσματικότητά τους. Αυτό είναι θετικό. Βέβαια, το να εφαρμόσουμε αυτή την τάση για να αντιμετωπίσουμε το υπερβολικό κόστος προβλέποντας μόνο 50% σε χρηματοδότηση, σε ένα ποσό που ήδη έχει μειωθεί, ε, είναι κατά τη γνώμη μου ασυνεπές από πολιτική άποψη, ούτε θα έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Γιατί στα υπόλοιπα ταμεία, στο ε, Κοινωνικό Ταμείο και στο ΦΕΝΤΕΡ έχουμε συγκεκριμένους στόχους που θα υλοποιηθούν. Στην περίπτωση όμως αυτή, όπου φαίνεται προφανές ε, έχουμε μεγάλη απομάκρυση, απόσταση, πελασιμότητα δυσχερή. Οπότε αυτό το κόστος το υπερβολικό στόχο θα έχει να μειώσει τις διαφορές. Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια διαφοροποίηση. Δεν βοηθάει στη σύγκληση, γιατί έτσι θα διευρύνεται το χάσμα και η, ανταγωνιστικότητα, η έλλειψη ανταγωνιστικότητας μεταξύ των περιοχών αυτών και της υπηρετικής Ευρώπης. Ένα άλλο σχόλιο που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι οποιαδήποτε στρατηγική για τις εξόχως απόκεντρε περιοχές θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ισορροπίες, τις ισορροπίες μεταξύ των παραδοσιακών μας δραστηριοτήτων και των ε, δραστηριοτήτων που στο μέλλον θα διαφοροποιηθούν και θα εξυγχρονιστούν. Επίσης, ε, άλλο σύγκληση και ποσά για το μετριασμό των δυσκολιών μας και άλλο ποσά που στόχο θα έχουν την προώθηση της μελλοντική μας ανάπτυξης. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί μπορεί να υπάρχουν κενά στη στρατηγική για τις εξόχως απόκαιτες περιοχές, αλλά δεν είναι όλοι οι στρατηγικές υφαλμένοι. Όντως, μερικές ε, περιοχές κατάφεραν να επιτύχουν σύγκληση πάνω από 15% τα τελευταία χρόνια, όπως η δική μου περιοχή. Κάτι που σημαίνει ότι οι πολιτικές αυτές είχαν και θετικά αποτελέσματα επιτόπου και αυτό θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε, να μην τα αλλάξουμε όλα άρδιν. Απλώς ε, θα προσθέσουμε κάποιους στόχους, θα βελτιώσουμε αυτό που ήδη υπάρχει, αλλά θα διαφυλάξουμε αυτό που απέδωσε καρπούς μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ, Λαμπέρ floor is yours. Yeah, ε, just... Ο λόγος εσάς. Ευχαριστώ για τα σχόλια. Πιστεύω ότι έχει σημασία σε αυτήν την περίοδο να δούμε το κείμενο με περισσότερες λεπτομέρειες. Τα πράγματα Φοβούμαι ότι έχουν αλλάξει από την εποχή που πρωτοσολήθηκαμε με το θέμα, διότι πλέον σωβεί μια κρίση. Διάφορα έργα περί απασχολησιμότητας κλπ. ολοκληρώθηκαν. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία άλλαξαν. Μιλάμε πια για την Ευρώπη του 2020. Μιλάμε για τη μεταβολή του κλίματος, την ενέργεια, την καινοτομία. Όλα αυτά συνάφε βεβαίω με την πολιτική συνοχή. Πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί λοιπόν στον εντοπισμό των ευκαιριών για την Γαλλική Βουιάννα για παράδειγμα. Ξέρω ότι το πρόγραμμα Γαλιλαίο έχει δραστηριότητε στην περιοχή. Από εκεί άλλωστε γίνονται και εκτοξεύσεις των γαλλικών πυράβλων. Ας δούμε λοιπόν ποιες είναι οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε αυτές τις περιοχές. Εδώ έχω ένα έντυπο που αφορά την ε, ψηφιακή ατζέντα όπου γίνεται λόγος για βιομηχανική πολιτική, απόδοση για εξειδικευμένες θέσεις εργασίας. Βλέπετε υπάρχει και εδώ μια πολιτική. Θέλω να πω με άλλα λόγια ότι υπάρχουν ευκαιρίε, αλλά πρέπει να μας πείτε κι εσείς για αυτές τις ευκαιρίες. Γιατί παράλληλα. Εξετάζουμε θέματα έρευνας και ανάπτυξης, αριστείας. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε υποδομές στα νέα κράτη-μέλη, τα οποία θα αποτελέσουν οχήματα ανάπτυξης. Βεβαίως, τα περισσότερα κονδύλια από τα παλιά προγράμματα πηγαίνουν σε παλιά κρατημέλη, αλλά κάνουμε πράγματα και για τις νέες περιοχές. Πιστεύω λοιπόν ότι κάτι παρόμοιο θα μπορούσε να γίνει και τις από κεντρές περιοχές. Στο πλαίσιο και της αντίληψης της ε, έκθεσης. Αναζητούμε λοιπόν νέες διαδικασίες. Τέλος, εγώ βεβαίω είμαι από την Ολλανδία. Βλέπω ότι ο κ. Ε, Σόλμπες μίλησε σοφά και συνετά. Πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση, να σκεφτούμε και τις ε, Ολλανδικές αντίληση των επόμενων χρόνων στο πλαίσιο του προπολογισμού και να έχουμε την αντίστοιχη υποστήριξη. Για να βοηθήσουμε ακριβώς αυτές τις περιοχές να κάνουν ένα βήμα προς τα εμπρός μεταξύ άλλων στον τομέα των επικοινωνιών. Ο Επίτροπος Πίβας ασχολείται με το θέμα εδώ και καιρό. Και με ενημέρωσε για τις προσπάθειες στην Ολλανδία. Αλλά αυτά πρέπει να γίνουν γρήγορα. Πιστεύω ότι χάρη και σε μια ορθή πολιτική επικοινωνία θα έχουμε πιο απτά αποτελέσματα. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Τεσέρο να κοιτάξει λοιπόν το μέλλον και να προχωρήσουμε. Ας ε, προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τις ευκαιρίες, να ανοίξουμε νέους δρόμους. Ας ε, δούμε την Ένωση σαν μια μεγάλη γειτονιά που χρειάζεται τέτοια πολιτική. Α υποστηρίξουμε λοιπόν τι νέε αυτέ προσπάθειε. Ευχαριστώ. Ε, Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπε ο Γιώχιμ Τσέλερ. Είπε ότι το πρόβλημα της Γαλλικής Γουιάννας έγκυται στο ότι λίγοι γνωρίζουν ότι υπάρχει αυτό το υπερπόντιο διαμέρισμα. Θα ήθελα να του πω ότι ε, είμαι στο Κοινοβούλιο αρκετά χρόνια, αλλά ορισμένα ζητήματα έχουν παραμείνει ακόμη ασαφή. Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε διευκρινήσει για διάφορα ζητήματα που βλέπω ότι επανέρχονται στη συζήτηση. Καταρχήν λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω. Μπορεί να οφείλεται στη δική μου άγνοια και αδαημοσύνη για τη συνθήκη. Μπορεί να γνωρίζω το συγκεκριμένο εδάφιο τη συνθήκη. Αλλά Ερωτώ, ποιος είναι ο ορισμός των εξόχως απόκεντρων περιοχών. Γιατί λέμε ότι μερικές ε, περιοχές λαμβάνουν το χαρακτηρισμό ή το καθεστώς ε, των εξόχως απόκεντρων περιοχών και άλλες περιοχές το χάνουν αυτό το καθεστώς. Δηλαδή δεν, δεν αρκούν κάποια γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για να δικαιούται κανείς το καθεστώς των εξόχων από περιοχών. Είναι σημαντικά αυτά τα σημεία γιατί το θέμα αν οι Ολλανδοί ε, υποβάλλουν την υποψηφιότητα του, νησού, του νησιού του ε, και θα προσθεθεί αρούμπα στι εξόχω απόκεντρε περιοχέ είναι ένα θέμα. Και άλλο θέμα είναι που η Γάλλη έχασε το Σαν Τελεμή. Να δούμε λοιπόν ποια κριτήρια εφαρμόζονται. Ε, υπάρχει και δεύτερο επίπεδο της συζήτησης ε, που αφορά τα νησιά, γιατί δεν είναι όλες εξόχως απόκεντρες περιοχές νησιά, ούτε κάθε νησί είναι και εξόχως απόκεντρη περιοχή. Σε λίγο θα ε, περάσουμε και στη συζήτηση ότι και τα νησιά δικαιούνται το καθεστώς των εξόχων απόκεντρων περιοχών μόνο και μόνο επειδή είναι νησιά. Ε, εδώ υπάρχει κάποια ανακρίβεια, γιατί άλλο νησιά και άλλο εξόχως απόκεντρες περιοχέ. Μπορεί μερικέ φορέ να υπάρχει επικάλυψη, αλλά όχι αυτόματα. Νομίζω ότι υπάρχουν και άλλα νησιά. Ήταν εκτό μικροφώνου δυστυχώ στο σχόλιο του κυρίου Τσέλερ. Ε, θα σα θερμοπαρακαλούσα να μου διαλευκάνετε αυτό το σημείο. Έχω και άλλη ερώτηση. Αν έχουμε εδώ να κάνουμε με συγκεκριμένες περιοχές, με, με συγκεκριμένο καθεστώς, και αυτές οι περιοχές ανήκουν σε συγκεκριμένες περιοχές, σημαίνει ότι υπάρχει και μία μονάδα που ασχολείται, ασχολείται με τις ε, εξόχως απόκεντες περιοχές. Η κυρία Άννα Πάουλα ασχολείται με αυτό. Δηλαδή ένα τμήμα ε, της ε, πολιτικής συνοχής αφορά τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και υπάρχει ειδική μονάδα που ασχολείται με το συντονισμό όλων των κοινοτικών πολιτικών για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Δηλαδή η πολιτική συνοχή συντονίζει και άλλες ε, κοινοτικές πολιτικές στον τομέα αυτό, ούτε και αυτό το γνωρίζω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο για τη συζήτηση, γιατί αν δεν ε, εξηγήσουμε όλα αυτά τα θέματα θα έχουμε προβλήματα. Άλλα προβλήματα αφορούν τις προκλήσεις των εξόχως απόκεντρο περιοχών. Ο κύριος Βανίστερόι μίλησε για τις ευκαιρίες, ε, τις νέες δυνατότητες που δίνουν οι νέες τεχνολογίες από τη μια πλευρά. Από την άλλη πλευρά έχουμε και δυσκολίες και δυσχέρειες στην πρόσβαση και υπάρχει το πρόβλημα της λειψιδρίας, ε, ε, της αξιοποίησης του ύδατος. Το είδαμε στη Μαδέρα στην επίσκεψη. Και το θέμα αυτό της άρδευσης ε, είναι πολύ δαπανηρό και συνιστά πρόβλημα ιδιαίτερα για τις εξόχως απόμακρες περιοχές. Πολλά προβλήματα και προκλήσεις απορρέουν από τη γεωγραφική τους θέση, αλλά υπάρχουν και κάποιες ευκαιρίες που οφείλονται επίση στη γεωγραφική θέση ή στη μείωση τη απόσταση ε, που δίνουν οι νέε τεχνολογίε. Και διαπίστωσα ότι μία από ένα από τα σημαντικότερα έσοδα του Λουξεμβούργου είναι οι δορυφορικέ συσκευέ. Όταν το έμαθα αυτό, διαπίστωσα ότι όλα είναι δυνατά τελικά. Το θέμα δεν είναι κανεί μεγάλο ή μικρό, πλούσιο ή φτωχό, αρκεί να έχει συγκεκριμένο είδο οικονομικέ δραστηριότητε. Λοιπόν, αυτέ τι διαλευκάσει θα ήθελα και τι διευκρινήσει για τις ερωτήσεις που σας έθεσα. Θα σας ήμουν ευγνώμων. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Μαρία. Ευχαριστώ. Θα ήθελα επί τη ευκαιρία να υποβάλω μια οριζόντια ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. <coughs> Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Σόλβες για την ε, πολύ οξυδερκή του έκθεση για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και κυρίως ε, να τον ευχαριστήσω για τις ελκυστικές και καινοτόμες προτάσεις ό,τι αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι περιοχές αυτές. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας μίλησε για την ποιότητα, την οριμότητα, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συμπληρωματικότητα, την κοινή λογική ε, εις βάρος των βασικών αρχών της αλληλεγγύης, της οικονομικής συνοχής, της κοινωνικής πολιτικής. Κύριε Σόλβε, θα ήθελα να σα υποβάλω μία ερώτηση. Ήσασταν κατά τη γνώμη μου από τους καλύτερους υπουργούς οικονομίας της Ισπανίας και με την πλούσια εμπειρία που έχετε. Σας ερωτώ πώς θα συνδυάζατε εσείς σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς την ανάγκη δημοσιονομικής πειθαρχία με την οικονομική και την κοινωνική συνοχή αλλά και την αλληλεγγύη. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Άρα λόγω στον καλεσμένο μας. Ε, η πόλεμος ε, μπορεί να διευκρινίσει ένα ερώτημα που αφορά την ένταξη στην κατηγορία των εξόχων από κέντρων περιοχών. Και από εκεί πέρα μπορείτε να απαντήσετε όπως θέλετε, να κατανοείτε το χρόνο όπως θέλετε με τον Επίτροπο. Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω πολύ σύντομα να το ξεκαθαρίσω γιατί ήταν εύλογη η ερώτηση. Να σας θυμίσω μερικά πράγματα από το παρελθόν. Δεν ήμουν εδώ. Ο κύριος Όλμπριχτ όμως μπορεί να θυμάται και ε, μπορεί να μην ξέρει το θεσμικό πλαίσιο, το νομικό πλαίσιο. Στη συνδίκη του Άμστερνταμ το 1999 ανέφερε τις εξόχως ε, από και τις περιοχές αναγνωρίζοντας την ανάγκη ειδική μεταχείρισής τους λόγω των γεωμορφολογικών περιορισμών που αντιμετωπίζουν. Στο άρθρο 299, οι περιοχές αυτές αναφέρονται. Το άρθρο αυτό είναι το άρθρο 349 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Πρόκειται για τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, Γουαδελούπη, Μαρτινίκα, Ουιάννα και οι νήσους Ριουνιών, στα οποία προσθέθηκαν δύο άλλα εδάφη για λόγους εσωτερικού γαλλικού δικαίου. Το Σαν Μαρτά και το Σαν Παρτελεμή με την ε, θέσπιση της ε, συνδίκη τη Λισαβόνα, τα δύο τελευταία εδάφια έγιναν ανεξάρτητες περιοχές και προσθέθηκαν στα υπερπόντια διαμερίσματα πλέον. Οι άλλε περιοχές, οι δύο αυτόνομε ε, περιοχέ περιοχές και Μαδέρα και τα Κανάρια και Καναρή νήσι συμπληρώνουν τον κατάλογο. Αυτά σύμφωνα με το άρθρο 349 τη συνθήκη τη Λισαβόνας. Υπάρχει όμω η δυνατότητα να προσαρμόζονται οι σχετικέ κοινωνικέ πολιτικές. Στο 355, στο άρθρο 355 όμως, υπάρχει μια διάταξη την οποία ονομάζουμε ρήτρα πασαρέλα με την εξή έννοια ότι η Γαλλία, η Ολλανδία και η Δανία δίνανται να ζητήσουν τροποποίηση του καθεστώτος μιας των περιοχών τους. Μην με ρωτάτε γιατί οι Πορτογαλοί, η οι Άγγλοι δεν έχουν το σχετικό δικαίωμα. Το καθαρό αποτέλεσμα πάντω είναι ότι η Γαλλία, η Ολλανδία και η Δανία έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τροποποίηση του καθεστώτο μια των περιοχών του. Στο πλαίσιο αυτό, ακριβώ, πρόκειψε το θέμα του Μαγιότ. Εάν δηλαδή οι κατοχώρε κρίνουν ότι μία από τι περιοχέ τους όπω είναι η Ολλανδική Συντήληση προκειμένου, πρέπει να κηρυχθούν εξόχως από την περιοχή, δίνεται να ζητήσουν, όχι στην Επιτροπή, αλλά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να γίνει η αλλαγή αυτή του καθεστώτος και αυτό κρίνεται βάση γνωμοδότηση τη Κομισιόν. Για το ΣΕΜΠΑΡΤΕΛΕΜΗ, λοιπόν, όπω είπα, ανακηρύχθηκε εξόχως από κεντρική περιοχή, απολάβοντας των σχετικών προνομίων όμω αλλάζει αυτή τη στιγμή το καθεστώ του. Γίνεται λέει, το αντίθετο, το αντίστροφο ακριβώ, Η Μαγιότ που είναι υπερπόνιο διαμέρισμα ζητά να γίνει εξόχω απόκεντρη περιοχή. Το Συμβούλιο πλέον θα κρίνει επί του και εμεί, η Κομισιόν αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε την γνωμοδότησή μα. Και επειδή ρωτήσατε και κάτι το οποίο αφορά τη δική μου μονάδα, την οποία έχω μεγάλη ε, υπερηφάνεια, και του Μονίκη βεβαίω, να πω γιατί το θέμα είναι, ανήκει στην Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο. Και εδώ υπάρχουν ιστορικοί λόγοι. Όταν έγινε μια αναδιάρθρωση τη Κομισιόν πριν από λίγα χρόνια και ο Επίτροπο Μπαρνιέ την εποχή εκείνη ήταν υπεύθυνο τη πολιτική συνοχή. στο πλαίσιο λοιπόν αυτή τη αναδιάρθρωση, μια μικρή μονάδα στη Γενική Γραμματεία τη Κομισιόν πέρασε στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής με συγκεκριμένη εντολή να συντονίσει όλες τις πολιτικές. Για να απαντήσω συγκεκριμένα λοιπόν στο ερώτημά σα, η μονάδα αυτή δεν ασχολείται μόνο με την πολιτική συνοχή. Προσπαθούμε κατά κάποιο τρόπο να υλοποιήσουμε το άρθρο 349, υπενθυμίζοντα τι ε, γενικέ διευθύνσει και μονάδε τη Κομισιόν ότι το άρθρο αυτό καταρχήν υφίσταται και ότι ο καταλόγος αλλάζει, υπάρχουν εξαιρεσει, ε, απαλλαγέ οι οποίε πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συγκεκριμένε περιπτώσει. Με συγχωρείτε, δεν θέλω να το συζητήσουμε από την αρχή. δεν θα πρέπει να λέμε λοιπόν εξόχως απόκεντρες περιοχέ, αλλά οι περιοχέ οι οποίε εντάσσονται ή απολάβουν του συγκεκριμένου καθεστώτο. Γιατί πρόκειται για καθεστώ και όχι για γεωγραφική ένδειξη. Είναι πρόκειται για χαρακτηρισμό. Στα αγγλικά τις λέμε outermost regions, πρόκειται για περιοχές που ανήκουν στα κράτη-μέλη, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που γεωγραφικά όμως βρίσκονται εκτός, Ευρωπαϊ... εκτός Ευρώπης, που απολαύουν όμως ε, όλου του κοινοτικού κεκτημένου. Όλο το κοινοτικό κεκτημένο εφαρμόζεται 100% εκτός από αυτά που προβλέπει, τις εξαιρέσεις, αν θέλετε, που προβλέπει το άρθρο 349. Ευχαριστώ. Εγώ έχω ένα γενικό σχόλιο. Ευελπιστώντας ότι θα απαντήσω στις ερωτήσεις. Αν κατάλαβα καλά, αυτό που είπε ο κύριος Τσέλερ είναι το εξής. Έχουμε τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, δεν τις αξιοποιήσαμε δεόντως, ώστε να γίνουν στο επίκεντρο της Ευρώπης. Μέχρι στιγμής θα το κάνουμε, ας το κάνουμε τώρα. Σύμφωνο απόλυτα. Ίσως ε, δεν δώσαμε αρκετή προσοχή μέχρι στιγμής. Ε, ε, μιλήσαμε για τη σύνδεση. Περισσότερο ασχοληθήκαμε με το πώς θα τη συνδέσουμε με την υπηρετική Ευρώπη παρά με τη, με τη γεωγραφική τους περιοχή, με τη γεωγραφική του ζώνη. Και όταν χρηματοδοτείται ένα πρόγραμμα σε μία γεωγραφική ζώνη, σε ένα υπερβόντιο διαμέρισμα, παρόλο που είναι το ίδιο σχέδιο, το ίδιο πρόγραμμα, υπόκειται σε διαφορετικά κριτήρια και μερικές φορές αντιφατικά και σε διαφορετική χρηματοδότηση. Γιατί ε, το ένα τμήμα του προγράμματος αφορά υπερβόντιο διαμέρισμα και άλλο τμήμα του προγράμματος ε, εξόχως απόκεντρη περιοχή. Αυτό που είναι σημαντικό στις εξόχως απόκεντρες περιοχές είναι να μην είναι στραμμένες ε, προς εμάς, αλλά να είναι σωστά ενταγμένε στην ευρύτερη ζώνη τους και στην ευρύτερη περιφέρειά τους. Έτσι θα αξιοποιηθεί καλύτερα το δυναμικό τους. Και φυσικά συμφωνώ μαζί σας ότι είναι τεράστιο το δυναμικό και οι δυνατότητες αυτών των περιοχών σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για παράδειγμα. Η προσφορά των εξόχως απόκεντρων περιοχών είναι τεράστια, ακόμη και από πειραματική άποψη. Το ίδιο ισχύει και για τις κλιματικές αλλαγές, το ίδιο ισχύει για την βιοπικιλότητα, για την αξιοποίηση των θαλασσών. Ε, στις εξόχως απόκεντρες περιοχές έχουμε λίγο, α, λιγότερο από το 50% των χωρικών υδάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ σημαντικά λοιπόν στοιχεία που χρήζουν τις δέουσες προσοχής. Ο κύριος Άλβες και εγκομιαστικά σχόλια έκανε, αλλά και επικρίσεις προς την έκθεση για την χαρακτήριζε υπερβολικά συγκεκριμένη. Ας ε, είμαστε σαφείς. Η έκθεση δεν αξιώνει να υπαγορεύσει τι θα πρέπει να γίνει. Το τι θα πρέπει να γίνει θα το κρίνουν το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκθεση δίνει το πρίσμα κάποιου εξωτερικού παρατηρητή που δίνει πληροφορίες για θέματα που θεωρεί σημαντικά και τα οποία αξίζει κανείς, στα οποία αξίζει κανείς να εγγύψει. Επίσης, όποια και είναι η απόφαση που θα ληφθεί, προτάθηκε να ε, μην λησμονεί αυτή η πρόταση της εξόχως κέντρες περιοχές. Πάντως δεν πρόκειται εγώ να σχολιάσω το συγκεκριμένο περιεχόμενο ενός τέτοιου σχεδίου, ούτε θα μιλήσω για χρηματοδότηση. Γιατί είπα ότι δεν περιορίστηκα από την ε, χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση είναι κάτι που θα έρθει αργότερα. Ε, προσπαθούμε να βρούμε μια καλύτερη ισορροπία. Ναι, μεν, αλλά το θέμα, το η έννοια των εξόχως απόκεντρων περιοχών δεν έχει ως αποκλειστικό στόχο την ισορροπία. Η ισορροπία ούτω ή άλλω είναι το ζητούμενο τη πολιτική συνοχή. Δεν περιορίζεται στι εξόχω απόκεντρε περιοχέ. Στι περιοχέ αυτέ αντιμετωπίζουμε ειδικά προβλήματα που δεν εμφανίζονται σε άλλε περιοχέ και που έχουν άλλη κατάσταση, ψηλότερο εισόδημα, αλλά παρόλα αυτά χρήζουν υποστήριξη όταν κανείς είναι πολύ απομακρυσμένος υφίσταται κάποιους φυσικούς περιορισμούς. Επίσης ο κατακαιρματισμός της αγοράς είναι ένα άλλο πρόβλημα γιατί δεν υπάρχουν απρόσκοπτες συγκοινωνίες και διασυνδέσεις με τις υπόλοιπες περιοχές. Ο κύριος Βανίστερ Ρόι μίλησε για κάτι πολύ σημαντικό. Ρώτησε τι γίνεται με το στόχο του 2020 και την κρίση. Η κρίση στις ε, υπεραπόμακρες περιοχές ήταν ε, ε, ολέθρια και η ανεργία έφτασε στο 30%, η ανεργία των νέων στο 50%. Παρόλο που οι κυβερνήσεις προσπάθησαν να, να βελτιώσουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το πρόβλημα των άνεργων νέων, των αποφύτων, είναι εμφανές σε όλη την Ευρώπη, αλλά πολύ περισσότερο στις εξόχως κεντρε περιοχές. Θα πρέπει όμω να αξιοποιήσουμε αυτό το δυναμικό, αυτό το ανθρώπινο κεφάλαιο και να ε, ενισχύσουμε τουλάχιστον την κινητικότητα. Αυτό το θέμα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Σίγουρα η παιδεία και η κινητικότητα είναι κρίσιμα στοιχεία. Επίσης, ε, οι νέες τεχνολογίες είναι θεμελιώδες σημείο και όπως είπα προηγουμένως, και η χρηματοδότηση είναι κέριο σημείο. Δηλαδή το ότι δεν έχουμε συστήματα προσαρμοσμένα στις περιοχές, συστήματα χρηματοδότησης, ε, δημιουργούν εξάρτηση αυτών από την υπηρετική Ευρώπη και τα κριτήρια που εφαρμόζονται δεν ισχύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν χρήζουν ανάλυση. Δεν ξέρω αν η λύση θα δοθεί από εκεί, αλλά τουλάχιστον μια διερεύνηση όλων αυτών των σημείων. Είναι αλήθεια ότι δεν πήγαμε στις Αντίλες, ε, Επισκεφτήκαμε όμως τις τότε οι ε, εξόχως απόκεντρες περιοχές. Στόχος μας ήταν ε, να εξετάσουμε την πολιτική της γειτονίας και επιμείναμε στο σημείο αυτό και στην ανάγκη όχι μόνο για τα υπερπόντια εδάφη και διαμερίσματα, για συγκεκριμένες ζώνες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν εντάσσονται στις ε, εξόχως απόκεντρες περιοχές, είπαμε ότι δεν θα πρέπει ε, να εστιαστεί μόνο σε αυτές οι πολιτική της γειτονίας, αλλά είναι κάτι ευρύτερο. Και η τελευταία ερώτηση, γιατί φαίνεται να πλανάτε μία αφιβολία. Μπορούν όλε όλες οι χώρες, αν είναι τις, δηλαδή, ε, η Δανία, η Γαλλία, η Ολλανδία να ζητήσουν χαρακτηρισμό τέτοιο εξόχω απόκεντρο περιοχών για οποιαδήποτε περιοχή. Όχι, έπρεπε αυτέ οι περιοχέ να είναι πολύ απομακρυσμένε, απομονωμένε. Και στο παρελθόν έτσι γινόταν η διάκριση, η διαφοροποίηση. Αλλά θα τα λέω από μνήμης, δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία. Και ένα άλλο θέμα που κατά τη γνώμη μου δεν έχει σχέση με την με τις από απόκεντρες περιοχές που δέθησε ένας ομιλητής. Πάντως η συζήτηση είναι ε, συναρπαστική για το πώς θα εξέλθουμε από την κρίση με, με πειθαρχία, με λιτότητα ή με εξάπλωση, με διεύρυνση. Αυτό είναι άσχετο με τις από απόκεντρες περιοχές, αλλά πιστεύω ότι αυτό θα εξαρτηθεί περισσότερο από την αντίληψη που έχει η αγορά για τη δυνατότητα μιας χώρας να χρεωθεί. Από αυτό εξαρτάται η έξοδο από την κρίση. Γιατί μπορεί κανεί να υιοθετήσει επεκτατική πολιτική, αλλά αν δεν βρει χρηματοδότε για αυτή, είναι καταδικασμένο προσπαθία Η προσωπική μου θέση είναι ότι εξαρτάται φυσικά από τη στάση τη κάθε χώρα, αλλά σε πολλέ χώρε το σημερινό περιθώριο ε, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι η λιτότητα, η εξυγίανση, ο περιορισμός και για το περιθώριο της πολιτικής ε, εξάπλωσης είναι να δοθεί προτεραιότητα στο δημόσιο χρέος στα στοιχεία που έχουν περισσότερη σημασία για την ανάπτυξη. Σε αυτά τα στοιχεία να δοθεί έμφαση και προτεραιότητα. Αυτά κατά τη γνώμη μου είναι κάποια γενικά στοιχεία που αφορούν τις δημοσιονομικές αποφάσεις και δεν αφορούν ιδιαίτερα τις από απόκεντρες περιοχές. Ευχαριστώ. Νούνο, θα ήθελες και εσύ να προσθέσεις κάτι, έχεις δικαίωμα να μιλήσεις τελευταίο ομιλητής, μια και είσαι ο Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν θα ήθελα να παρατείνω τη συζήτηση. Δύο λόγια μου μόνο. Θα ήθελα να πω ότι βρισκόμαστε στην αφετηρία αυτής της συζήτησης γιατί σίγουρα η κέρη είναι χαλεπή, πολλά σημεία θα πρέπει να συζητήσουμε και να διαπραγματευτούμε, αλλά νομίζω ότι είναι και η ώρα να περάσουμε από τα λόγια στα έργα. Έχουμε πολλά στοιχεία να αναλύσουμε και ελπίζω ότι η Επιτροπή μας με όλες αυτές τις ε, συνεισφορές και τις παρατηρήσεις ε, να δώσει τον αρκτήριο Λάκτης μας αυτή τη συζήτηση και έχουμε και την ανακοίνωση που περιμένουμε του χρόνου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Προσβλέπουμε σε αγαστή συνεργασία με τη μονάδα της κυρίας Αναπάουλα ε, και της Γενικής Διεύθυνσης Ρέτζιου. Ελπίζουμε να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο και να προστατήσει η Γενική Διεύθυνση αυτή θέτοντα στο επίκεντρο τη εξόχω απόκεντρε περιοχές και φέροντα αίσιο πέρα τις σχετικέ προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που ήρθατε και συμμετείχατε στη συζήτηση. Και εγώ να ευχαριστήσω με του δύο καλεσμένου μας. Πιστεύω ότι στην έκθεση θα διαβάσουμε πολλά, τα οποία θα μας εμπνεύσουν για τη δική μας έκθεση και τις συστάσεις μας. Θεωρούμε ότι η Γενική Διεύθυνση δείχνει το δρόμο με υπευθυνότητα και στον τομέα των εξόχως αποκεντρωμένων απόκεντρων με περιοχών. έρθει τη ώρα και για τις διαπραγματεύσεις θα μας πείτε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες προκλήσεις. Πέτρο, έχεις δίκιο. Πρέπει να προσέξουμε με τις δαπάνε. Να δούμε ποιες δαπάνες οδηγούν σε ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε εποχές που δίδει χρημάτων. Η πρόκληση είναι αυτή ακριβώ να χρησιμοποιήσουμε την πολιτική συνοχή εκεί που οι πόροι λείπουν, ως, ως καταλήτη, ως μοχλό, αν θέλετε, για να προσελκύσουμε και άλλα επιπλέον κεφάλαια και να προκαλέσουμε ανάπτυξη. Αυτό είναι η πρόκληση. Ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Uh, dear colleagues, uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, ένα μεγάλο θέμα μας έχει μείνει στη μερική διάταξη και ένα μικρό. Ε, δώστε μου όμως ε, δύο λεπτά για να σας ενημερώσω για τις αποφάσεις που λήθησαν εχθές από τους συντονιστές, διότι έχουμε μοιράσει αρκετές νομοδοτήσεις και εκθέσεις. Ενημερώνω ότι ο κανονισμός για το Ταμείο, το EGF, προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση πάει σε σοσιαλιστέ και φιλελεύθερου. και, ε, ε, ε, και δημοκράτε, με συγχωρείτε ή το πακέτο για τα αγροτικά ο σχετικό κανονισμό για τι άμεσε πληρωμές στους αγρότε που πηγαίνει στους πράσινου, μία άλλη στο ECR και ο κανονισμό για την κοινή οργάνωση αγοράς στην ΚΟΕ Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκό Ταμείο Γεωργίας Αγροτική ε, Ανάπτυξης ε, στους πράσινους και ο κανονισμός ε, Κοινοβουλίου Συμβουλίου για την διαχείριση χρηματοδότησης γεωργικής πολιτικής στην ΑΛΔΕ, κανονισμός για την εφαρμογή των αμέσων πληρωμών στους αγρότες για το 2013 επίσης ΑΛΔΕ, Connecting Europe, μηχανισμός Connecting Europe, στο ΕΛΚ, κανονισμό για τις ενεργειακέ υποδομέ στου ε, σοσιαλιστές, τηλεπικοινωνίε ALDE και τα TEN, τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών στην ECR. Μη νομοθετικέ νομοθετήσει για την μεταρρύθμιση της κοινή ελευθερικής πολιτική στο ΕΛΚ, ελκυστικότητα επενδύσεων ECR, διαχείριση ποιότητα ευρωπαϊκών στατιστικών στο ΕΛΚ και μικρής κλίμακας αλία στους πράσινους. Να σε ενημερώσω επίσης ότι ζητήσαμε από την γραμματεία να εξετάσει όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν πρακτικά όσον αφορά την συνεργαστία της Γενικής Διεύθυνσης ε, Ρέτζι με τις επιτροπές που έχουν συναφεί ενδιαφέροντα. Όσον αφορά την νομική γνώμη για το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, σα ενημερώνω ότι λάβαμε από την νομική μας υπηρεσία την πληροφορία ότι ευθυγραμμίζεται με τα όσα λέμε τα τελευταία χρόνια, ότι δηλαδή πρέπει να υπόκειται στην τακτική νομοθετική διαδικασία και όχι αυτό το οποίο προτείνει η Κομισιόν με κατεξουδότηση δηλαδή πράξη. Θα ενημερώσω τον Επιτροπό Χάν με της αποφασιός μας, αν δεν έχετε φυσικά αντίρρηση εδώ. Και με αυτά, να περάσουμε στο επόμενο σημείο στην ημερησία διάταξη. Κόβατσεφ, για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 14-20. Παρακαλώ. τη συνάδελφη θα μιλήσω βουλγαρικά. τέλος του έτους η Κομισιόν υπέβαλε τις σχετικές προτάσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Πώς θα έχουμε περισσότερη Ευρώπη με τα ίδια κονδύλια. Ο διάλογος αυτή τη στιγμή είναι μεταξύ αυτών που θέλουν περισσότερη Ευρώπη και αυτών που θέλουν να συρρυκνώσουν τον προπολογισμό. Ο πρώτος γύρος συζήτηση έλαβε χώρα. Και πρέπει να προωθήσουμε την περιφερειακή πολιτική διότι καταρχήν πρέπει να δούμε τον δημοσιονομικό κανονισμό και θα προχωρήσω κατευθείαν εις τα ε, συμπεράσματα που ασχολούνται με δύο θέματα, την ευρωπαϊκή συνεργασία και την εδαφική κατανομή. Ε, έχουν προταθεί 360 ε, δις τα οποία θα αναφερθούν στην ανάπτυξη και σε την δημιουργία θέσεων εργασίας θα υπάρξει ένα ποσό 11,7 δις το οποίο ε, θα αποδοθεί σε ε, διασυνοριακή συνεργασία και ε, διεθνική όπως και διαπεριφερειακή. Έχουμε προβλέψει να υπάρξουν ε, μία μείωση κατά 2,5%. Θα χρειαστεί επαναχάραξη ορίων περιοχών και δημόρφωση νέων κατηγοριών. Λαμβάνομαι υπόψη του ΑΕΠ ε, με μια νέα κατηγορία η οποία θα είναι μεταξύ 75% και 90% του μέσου κοινωτικού όρου. Έτσι θα καθοριστούν και τα όρια, τα ανώτερα όρια χρηματοδότησης για κάθε κατηγορία. Αυτά έχουν ως εξής. 75% στην πρώην κατηγορία σύγκλησης, 60% στις ε, περιοχές μετάβασης και 50% σε όλες τις άλλες περιοχές. Έχουμε επίσης τον κανόνα νη συν 2 που θα ισχύσει σε όλους τους τομείς εκτός από ένα των οποίο θα ισχύσει το νησιν 3. Το 50% αποτελεί ένα αποθεματικό το οποίο θα απελευθερωθεί στην αρτήση αποτελεσμάτων. Έχουμε εισαγάγει επίσης τη λεγόμενη θεματική συγκέντρωση των κονδυλίων. Υπάρχουν υποχρεωτικέ προτεραιότητε στην έρευνα και τεχνολογία καθώ και στην καινοτομία. τρει νέε κατευθύνσει. Ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και χαμηλέ εκπομπέ. Αυτό σημαίνει ότι οι λιγότερο ανεπτυγμένε περιοχέ θα χρειαστεί να επενδύσουν τουλάχιστον 50% των κονδυλίων που θα λάβουν σε αυτού του τομεί. Για τι περιοχέ μετάβαση, το ποστό αυτό είναι 50%, και τις πιο ανεπτυγμένες 80%. Όσον αφορά την υποχρεωτική πρωτοβουλία για, τις, τη μείωση των εκπομπών, οι περιοχές πρέπει να επενδύσουν μεταξύ 6 και 20% στον τομέα αυτών, ανάλογα το σε ποια κατηγορία ανήκουν. Τουλάχιστον επίσης 5% του ΕΤΠΑ πρέπει να δαπανηθεί σε εθνικό επίπεδο για την βιώσιμη ανάπτυξη των αστικών περιοχών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ταμείο Συνοχής θα επικεντρωθεί στις περιοχές με ΑΕΠ κάτω του 90% του κοινωτικού μεσουόρου. Έχουμε όμως και το μηχανισμό Connecting Europe, ο οποίος υποστηρίζει μεγάλα έργα υποδομής, το οποίο θα πρικοδοτηθεί με 50 δισεκατομμύρια, τα 10 είναι από το Ταμείο Συνοχή και αυτά θα δοθούν σε μεγάλα ευρωπαϊκά ε, έργα ανεξαρτήτως χώρα. Ο σχετικό διάλογος, η σχετική συζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει και είμαι σίγουρο ότι θα συνεχιστεί μέχρι να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Τα έργα του ΕΚΤ, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, θα υποστηριχθούν με εθνικέ χρηματοδοτήσει. Ε, τουλάχιστον 25% για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, 40% για τη μετάβαση και 50% για τις πιο ανεπτυγμένες περιοχές σε κάθε κράτος μέλος. Αυτή είναι η φιλοσοφία των νέων προτάσεων. Έχουμε και μια διαχειριστική, διαδικαστική δημορφία. Ο αυξημένο ε, ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά από την θέσπιση τη ε, συνδίκη τη Λισαβόνα δυστυχώ ε, δεν αποτυπώνεται στην ε, διαδικασία συνένεσης που προβλέπει η Λισαβόνα. Έτσι δεν επιτρέπεται ακόμη στο Κοινοβούλιο να έχει μεγαλύτερο λόγο στα σχετικά. Οι υπόψεις τη Επιτροπή του ΕΤΠΑ θα εξαρτηθούν και από τι δικέ σα ε, απόψει και την Επιτροπή Προπολογισμών. Να σας ενημερώσω ότι η Καθήλυνα Αρμόδια Επιτροπή Προϋπολογισμών προσπαθεί να αποκτήσει σημαντικότερο ρόλο εξ ονόματο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πράγματα αυτά και όχι μόνο απλώς να εγκρίνει να απορρίπτει προτάσεις. Θα μπορεί να συμμετέχει στη συζήτηση διαμεσών εκθέσεων για παράδειγμα. Όμως στη φάση αυτή, αυτή είναι η κατάσταση όπως σας την περιέγραψα, είμαι στη διαθεσή σας για σχόλια και ερωτήσει. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αυτή τη φάση μπορούμε μόνο να πούμε ένα ναι ή ένα όχι. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Σταυρακάκη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν είναι σημαντικό ότι στην ανακοίνωση της Επιτροπής προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020 αναγνωρίζεται ότι η πολιτική συνοχής δεν είναι απλά μια πολιτική αλληλεγγύης που στηρίζει τις πιο αδύναμες περιφέρειες. Αποτελεί επιπλέον μια πολιτική επενδύσεων η οποία είναι απολύτως απαραίτητη για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, η προστιθέμενη αξία της αποδεικνύεται από το γεγονός ότι πολλές επενδύσεις στον τομέα της ανάπτυξης και της απασχόλησης δεν θα είχαν γίνει χωρίς τη συνδρομή της πολιτικής συνοχής. Αναφορικά τώρα με την πρόταση κανονισμού, η οποία αποτελεί την ομοθετική μεταφορά αυτής της ανακοίνωσης, θα ήθελα να σταθώ σε κάποια σημεία τα οποία στηρίζονται με το έργο της Επιτροπής μας και θεωρώ ότι είναι πρωταρχικής για εμάς σημασίας. Καταρχήν, αναφορικά με τα κονδύλια που κατανέμονται στην πολιτική συνοχή για την επόμενη προγραμματική περίοδο, θα ήθελα να πω ότι δεν είμαστε απολύτω ικανοποιημένοι. Όπω όλοι γνωρίζετε, πάγιο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν η διατήρηση του ύψου των κονδυλίων, τουλάχιστον στο ύψο τη τρέχουσα περίοδου. Η Επιτροπή όμω δεν διασφαλίζει με την πρότασή τη αυτά τα ποσά. Κατά δεύτερον, καλωσορίζουμε τη δυνατότητα για τη μεταφορά των χορηγήσεων που δεν χρησιμοποιήθηκαν το 2014 στα επόμενα έτη, σε περίπτωση που κάποια, κάποια προγράμματα των τομέων το Ταμείο της Πολιτικής Συνοχής υιοθετηθούν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2014. Θα ήθελα ωστόσο να τονίσω εδώ τη σημασία της έγκαιρης έγκρισης τόσο των κανονισμών των ταμείων όσων και των συμβάσεων εταιρική σχέση και των επιχειρησιακών προγραμμάτων, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η υλοποίηση τη νέα γενιά προγραμμάτων θα αρχίσει το συντομότερο δυνατόν. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθούν πολλά προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την έναρξη κάθε προγραμματική περίοδου. Αυτό πρέπει να αποτελεί κύρια προτεραιότητα στο έργο μας στους επόμενους μήνες. Επίσης, πρωταρχική σημασία είναι η ανάγκη διασφάλισης της σωστής ισορροπίας μεταξύ από τη μία της αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας και της προβλεψιμότητας των δαπανών και από την άλλη τη ευελιξίας που απαιτείται ώστε να μπορεί η Ένωση να αντιμετωπίσει τις απρόβλεπτες προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό καλωσορίζουμε γενικότερα τις διατάξεις για τα μέσα ευελιξίας και κυρίω την αναγνώριση του Ταμείου αλληλεγγύης. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω τις επιφυλάξεις μας αναφορικά με το μηχανισμό συνδέοντας την Ευρώπη με το γεγονός ότι υπάγεται στον προπολογισμό της πολιτικής συνοχής. Όπως έχει ξεκαθαριστεί, η διαχείριση του νέου μηχανισμού θα γίνεται κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την βάση της πολιτικής συνοχής που είναι η επιμερισμένη διαχείριση. Επιπλέον, ένα ποσό ύψους 10 δις ευρώ προερχόμενο από το Ταμείο Συνοχής προβλέπεται ότι θα κατανέμεται για την υλοποίηση έργων του μηχανισμού συνδέοντα την Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώ θα συνδυαστεί και πώ θα λειτουργήσει στην πράξη κεντρική με την επιμερισμένη διαχείριση στο πλαίσιο του ίδιου μηχανισμού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω απλώς μία ερώτηση σχετικά με τη διαδικασία. Δεν ήξερα καν ότι πρέπει όχι μόνο να ψηφίσουμε το δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και όλα αυτά τα δύσκολα θέματα των ποσοστώσεων, των κατανομών. Βέβαια ξέρω ότι υπάρχει η διαδικασία ε, συμμετοχής ε, και συναποφάσεως αλλά αν ε, ε, δεν έχει το δικαίωμα εμβάσεως στο νομοθετικό έργο η Ολομέλεια τότε δεν ξέρω πώς θα προχωρήσουμε δηλαδή ε, ποιες είναι οι δυνατότητες μας αν επηρεάζουμε το νομοθετικό πακέτο ή όχι Κάπως τα έχω χαμένα αυτή τη στιγμή, να σας πω την αλήθεια δηλαδή. Ε, ο κύριος Τσέλερ και μπορεί να απαντήσει αν θέλει. Ευχαριστώ. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Διότι εδώ όντως βρισκόμαστε κάπου δέσμοι. Δηλαδή μας πιαστήκαμε σε μία παγίδα, είμαστε σαν το σκύλο που τρώει την ουρά του και ε, βάσει των απόψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε κάπως ε, παγιδευτεί στο δημοσιονομικό πλαίσιο οπότε αυτά που είπαμε χθες και σήμερα και τα αμφισβητήσαμε θα θεωρηθούν ότι τα έχουμε υιοθετήσει και δεν χρειάζεται πλέον να το συζητήσουμε ούτε για ποσοστώσεις, ούτε για συνδυάσεις. Ε, ε, για συνδυασμούς διότι δεν πρόκειται να μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα. Οπότε είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε επιγόντως με την Δημοσιονομική Επιτροπή διότι διαφορετικά δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε και να έχουμε μία βάση συζητήσεως για τις, ε, τους κανονισμούς. Ως εκ τούτου πρέπει να ενεργήσουμε πάρα πολύ γρήγορα. ευχαριστώ. Αντιλαμβάνομαι ότι ο κύριος Κάλφιν είναι εδώ, οπότε είναι ένας από τους δύο εισηγητές στην Επιτροπή Προϋπολογισμού, ο άλλος είναι ο Ράιμερ Μπέγκε, αλλά μπορούμε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κάλφιν, διότι εφόσον έχουν γίνει οι αρχικές παρατηρήσεις μπορείτε και εσείς να σχολιάσετε. Μπορείτε να του επαναλάβετε την ερώτησή σας αν θέλετε κυρία Κρέλ. Με συγχωρείτε, τότε θα επαναλάβω πάλι την ερώτησή μου, διότι ουσιαστικά δεν καταλάβαμε στην Επιτροπή ποια θα είναι η διαδικασία. Η έκθεση που καταρτίστηκε από την Επιτροπή Προπολογισμού δεν ακολουθεί τη διαδικασία συναπόφασης και μόλις ενημερώθηκα ότι δεν αναφέρεται μόνο στο συνολικό πλαίσιο για, την, ε, ε, για τα κεφάλαια συνοχές αλλά και ε, για όλες τις λεπτομέρειες, τις ποσοστώσεις, τις κατανομές, δηλαδή όλο το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θέλαμε εμείς να αποφασίσουμε. Και αμφισβητείται αν πρέπει να υπάρξει 20% ε, για την ενεργειακή αποδοτικότητα ή ένα ποσοστό για τις ε, λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Αν όντως προχωρήσουμε έτσι, σημαίνει ότι δεν χρειάζεται πια να προβούμε σε νομοθετική εργασία. Έτσι είναι ή είναι διαφορετική η κατάσταση, μπορείτε να μου απαντήσετε. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν ε, ζητώ συγγνώμη που έφτασα κάπω ε, καθυστερημένα, αλλά συμμετείχα στο τριμερή διάλογο για τον προπολογισμό του επόμενου έτου. Θα είμαι σχεδόν επιγραμματικό. Θα προσπαθήσω να απαντήσω και στην ερώτηση τη Κωνσταντζα. Προ το παρόν είναι σαφέστατη η εντολή ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και περιορίζεται από αυτά που ψηφίζαμε στην έκθεση Γκαρίγκα της Επιτροπής Σούρα. Επίσης έχουμε δύο εκθέσεις ίδιας πρωτοβουλίας για την συνοχή και την πολιτική γεωργίας. Προς το παρόν έτσι οριοθετείται η σαφέστατη εντολή που ενέκρινε για μας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιπλέον έχουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ε, βρισκόμαστε σε πολύ πρόωρο στάδιο της συζήτησης στο Συμβούλιο. Κατά πάσα πιθανότητα είναι ότι στις διαπραγματεύσεις θα μας προσκαλέσει ευγενικά η Πολωνική Προεδρία. Πριν και μετά κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων έχουμε briefing και την briefing. Ε, το επόμενο Συμβούλιο θα γίνει στις 5 Δεκεμβρίου. Είχαμε και πρόσφατα ένα. Και η στην τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων θα εξεταστεί κοινή γεωρική πολιτική και η πολιτική συνοχής. Στο Συμβούλιο της 5ης Δεκεμβρίου θα συζητηθεί το θέμα των ίδιων πόρων. Ουσιαστικά στο Συμβούλιο γίνεται μια απλή ανταλλαγή απόψεων. Δεν θα έλεγα καν ότι το Συμβούλιο προσπαθεί να συγκροτήσει μια θέση. Προς το παρόν εμείς έχουμε θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ανταλλαγή απόψεων ε, στο Συμβούλιο. Επίσημα δηλαδή οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο δεν έχουν ξεκινήσει. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, αυτό που ακούσαμε από την Πολωνική Προεδρία είναι το επόμενο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της 5ης Δεκεμβρίου θα είναι το τελευταίο και εκεί θα γίνει μία ανταλλαγή απόψεων για το θέμα των ιδίων πόρων. Στη συνέχεια, η Δανική Προεδρία φιλοδοξεί να, καταλή, να επιτύχει συμφωνία για την διαπραγματευτική εντολή, όπως τη χαρακτηρίζουν. Δηλαδή το επόμενο εξάμεινο, στη διάρκεια της Ιδανικής Προεδρίας, πολύ πιθανό θα καταλήξει το Συμβούλιο σε μια θέση με τους βασικούς άξονες, χωρίς ποσά μάλλον. Οπότε θα, θα διαπιστώσουμε πού συμφωνούμε, πού διαφωνούμε και πού δεν συμφωνούμε ακόμη, αλλά πολύ πιθανό να συμφωνήσουμε στο μέλλον. Αυτή θα είναι η βάση για τις διαπραγματεύσεις. Αλλά προς το παρόν ε, τίποτα παραπάνω δεν περιμένουμε από τη Δανική Προεδρία. Αυτές μέχρι εκεί φτάνουν οι φιλοδοξίες της. Προς το παρόν πάντως και πριν ξεκινήσουμε τις ουσιαστικές α, τυπικές επίσημες διαπραγματεύσεις, δεν πρόκειται να παρεκκλίνουμε από την εντολή που, έχουμε, που μας έχει αναθέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό ψηφίσαμε. Ούτε ε, ε, προς το παρόν έχουμε ανάγκη παρέκκλησης. Πρώτα θα ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις και μετά θα πρέπει να συμφωνήσουμε. Υπάρχει μια διαδικασία που αποφάσισε η διάσκεψη των Προέδρων και θα συνεννοηθούμε για το πώς θα συμπεριλάβουμε όλες τις επιτροπές στη συζήτηση. Ίσως ε, θα δημιουργήσουμε μια ομάδα επαφής και με, τον, με τους ώστε να ενημερώνονται συνεχώς όλες οι επιτροπές για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Και στη συνέχεια για, να δούμε πού υπάρχουν διαφορές σε σχέση ε, με την, επιτροπή, την έκθεση Επιτροπή ΣΟΥΡ και τη θέση του Συμβουλίου. Εμείς έτσι βλέπουμε την συνέχιση της διαδικασίας. Πάντως, στο πρώτο Συμβουλίο Γενικών Υποθέσεων που έγινε πριν από δύο εβδομάδες, διαπιστώσαμε που υπάρχουν διαφορές μεταξύ της δική μα έκθεση και της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρόβλημα είναι ότι η Επιτροπή προβλέπει μείωση των διαρθωτικών ταμείων και αύξηση του ταμείου μεταφορών. Και ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να, συμπεριλάβει το χρηματοδοτικό μέσο συνδέοντας στην Ευρώπη στο Ταμείο Συνοχής, αλλάζοντας τη δομή του προϋπολογισμού και καθιστώντας πιο ελαστική τη μεταφορά των κονδυλίων. Προσθήκης ή αφαίρεσης, στην περισσότερες περιπτώσεις αφαίρεσης κονδυλίων. Δεν ξέρω, θα συμφωνήσουμε με αυτή τη διαφορετική δομή που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, το χρηματοδοτικό μέσο συνδέοντας την Ευρώπη θα συμφωνούμε ότι εντάσσεται στην πολιτική συνοχή. Κατά τη γνώμη μου, ε, δεν εντάσσεται. Χθε παρουσιάστηκε αυτό το μέσο συνδέοντα την Ευρώπη στην Επιτροπή Ήτρε. Νομίζω ότι περισσότερο αφορά σχεδόν εμπορικά σχέδια. Νομίζω ότι για αυτό το λόγο έχει ε, προταθεί. Για προγράμματα που είναι κοντά στην εμπορική χρηματοδότηση. Δεν έχει βρεθεί ακόμη, αλλά δεν θα είναι επιχορηγήσει στα κονδύλια αυτού του χρηματοδοτικού μέσου. Το πρόβλημα είναι τα σχέδια αυτά όντως θα στραφούν σε περιοχές που χρειάζονται κάποια βοήθεια ή το σύνδετο στην Ευρώπη θα είναι κάτι ξεχωριστό και δεν θα βοηθά στην ενίσχυση της συνοχής των περιοφερειών. Επίσης, συμφωνήσαμε για το ενδιάμεσο καθεστώς των ε, περιοχών στο Κοινοβούλιο. Και την ίδια πρόταση την είδαμε και στη, στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά δεν ξέρουμε θα, αν θα προταθούν συμπληρωματικά κονδύλια ή θα εξαχθούν από τα κονδύλια της συνοχής. Μέχρι στιγμής ε, διαπιστώσαμε ότι ενδιάμεσα σε αυτές τις περιοχές, οι μεταβατικές περιοχές θα συμπεριληφθούν στα ποσά που χρησιμοποιήθηκαν μέχρι τώρα στο κονδύλιο της συνοχής. Οπότε έτσι μειώνονται συνολικά τα κονδύλια που απευθύνονται στις φτωχότερες περιοχές, τα κονδύλια της συνοχής. Αυτές είναι οι διαφορές μεταξύ της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της δικής μας πρότασης. Τώρα, αυτή είναι η μεθοδολογία. Όταν είπα ότι υπάρχει σαφή μείωση του Ταμείου Συνοχή, των κονδυλίων συνοχή, με βάση την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και αυτό εξαρτάται από τη βάση υπολογισμού που χρησιμοποιούμε για να καταμετρήσουμε αυτή τη μείωση. Η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ το παρόν είναι οι τρέχουσε τιμέ του 2011. Εμείς προτείνουμε να ληφθούν υπόψη οι στη τιμές του 2013, που είναι το τελευταίο έτος εφαρμογής του ισχύοντος πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου. Και έχουμε εξήγηση για, το, για, το, για την πρόταση αυτό, γιατί αν λάβουμε ω σημείο αναφορά το 2011 θα έχουμε μείωση ε, στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, μείωση της τάξης του 5,3% των, ε, των κονδύλιων συνοχής. Ενώ αν λάβουμε σημείο αναφοράς ε, το 2013 έχουμε 8,4% μείωση των κονδυλίων συνοχή σε σύγκριση με το ισχύον πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτή, αυτές είναι οι προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς εμένουμε στο ψήφισμα και την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα δούμε τι, τι θέση θα διαμορφώσει το Συμβούλιο. Πάντως, επαναλαμβάνω, ενδιάμεσες ή μεταβατικές περιοχές, πώς θα συνδέσουμε τις μεταφορές και το συνδέοντα στην Ευρώπη με την πολιτική συνοχής και η ελαστικότητα της πολιτικής συνοχής με διαφορετική ονομασία, με το ονομασία διαφόρων σημείων του προϋπολογισμού και τέλος ποιο έτος θα είναι το σημείο αναφοράς. για το αν θα έχουμε μείωση και τι επίπεδο θα είναι αυτή η μείωση ανάλογα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για συγκεκριμένα έτος αναφοράς. Ευχαριστώ κυρία Έρμς. Ευχαριστώ. Ε, είμαι σκεπτική ε, και επιφυλακτική όταν ακούω όλα αυτά ότι ε, μιλάμε για περί πολιτική συνοχής γιατί πιστεύω ότι είναι ασταθές το έδαφος το οποίο κινούμεθα τώρα και θα πρέπει να έχουμε τις αντιδράσεις των διαφόρων κρατών μελών. Ο παραδείγματος χάρη από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο στη Γερμανία λέγεται ότι αν το σύνολο του προϋπολογισμού ε, ε, ε, ξεπεράσει το ένα δις δεν θα ακολουθήσουμε. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι είναι σημαντικοί και μπορώ απλώς να ελπίζω ότι θα υπάρξει μία συμφωνία με τις ε, κατά τρόπον ώστε να συζητάμε συγκρίσιμα στοιχεία και να μην συζητάμε για πράγματα που δεν συνάδουν πλέον με το δημοσιονομικό πλαίσιο διότι διαφορετικά θα πρέπει να συζητήσουμε τους μεμονωμένους τομείς να δούμε τι προχωράει, τι όχι ε, και ε, θα ήθελα να το τονίσω διότι ε, ε, θεωρώ ότι είναι λίγο συγκεχημένο. Πρέπει ίσως να κάνουμε μία κοινή συνεδρίαση με τους υπευθύνους του προϋπολογισμού. Δεν θέλω να πω ότι πρέπει να κινητοποιηθούμε, αλλά νομίζω ότι για τη συνοχή αυτά τα στοιχεία είναι το, ο άγνωστος χ. Ευχαριστώ. Έχω να κάνω και μία δεύτερη ερώτηση. Αντιλαμβάνουμε ότι υπάρχει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η δικιά μας, και έχουμε ένα πηλίκον ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 360 ε, δις ε, ευρώ που κατανέμονται για πιο καλά ε, για καλύτερα ανεπτυγμένες περιοχές, ε, ενδιάμεσες περιοχές, ε, διασυνοριακή συνεργασία και ούτω καθεξής. Τότε, όπως και στο παρελθόν, θα μπορούσαμε όλα αυτά να τα βάλουμε σε αγγίλες και όταν θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για το μέσο πρόθεσμο δημοσιονομικό πρόγραμμα να τα διευκρινίσουμε. Αλλά ελέγχθη ότι επιπλέον υπάρχουν ε, στην πρόταση αυτή και άλλα πολύ σημαντικά για το δημοσιονομικό πλαίσιο 80% πρέπει ε, να χρησιμοποιηθεί στις πιο ε, ανεπτυγμένες περιοχές ε, για συγκεκριμένα προγράμματα, 20% για ενεργειακά προγράμματα στην ενδιάμεση κατηγορία θα πάει ένα ποσοστό στις πιο ανεπτυγμένες κάτι άλλο. Υπάρχουν δηλαδή ποσοστά τα οποία αξιολογούνται πάρα πολύ κρίσιμα. Αλλά κατά τη γνώση μας δεν ε, είναι θέματα ε, δημοσιονομικά αλλά είναι θέματα νομοθετικά ε, του νομοθετικού πακέτου. Ποια είναι η διαδικασία. Εσείς κάντε την επιλογή. Πρέπει να διαπραγματευτούμε επί του παραλίλου. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μήπως σε παρακαλώ μπορείς να μου τα σχολιάσεις όλα αυτά για να καταλάβω πού βρισκόμαστε. δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν παράλληλες διαπραγματεύσει Άλλωστε με ποιον, διότι το Συμβουλίο έχει τη δεδομένη θέση. Μιλάμε όμω για το εξή. Να σε εξηγήσω τι γενικέ δομέ Στην έκθεση του Κοινοβουλίου λέει ότι δεν χρειαζόμαστε λιγότερα κονδύλια το αντίθετο σε σχέση με το παρόν δημοσιονομικό πλαίσιο. Και από εκεί πέρα συζητάμε. Το Connecting Europe περιλαμβάνεται ή όχι ε, κινούμαστε με βάση τις τιμές 2011 ή όχι. Η Κομισιόν θα πει τότε ότι έχουμε αύξηση στις ονομαστικές τιμές 2,4. Ακόμα όμως και αν τα δούμε διαφορετικά τα πράγματα, πάλι μιλάμε για μείωση περίπου 5%. Αυτά είναι τα νούμερα. Να δούμε τώρα πώς το Συμβούλιο θα διαμορφώσει τη θέση του. Πριν να γίνει αυτό δεν μπορούμε να έχουμε καμία διαπραγμάτευση. Ακούμε διάφορα για την εσωτερική διαπραγμάτευση στο Συμβούλιο. Ξέρουμε ότι στο τελευταίο Συμβούλιο η πρόταση ήταν να αλλάξει η μέθοδος της διαπραγματεύσης, να συμφωνήσουμε πρώτα για τα νούμερα και μετά να δούμε για την κατανομή και τα άλλα. Μετά η Πολωνική Προεδρία υιοθέτησε την σωστή κατά μου προσέγγιση. Να μελετήσουμε, να αποφασίσουμε το περιεχόμενο της ε, στατικής 2020 ε, και μετά να δούμε τα νούμερα. Το Συμβούλιο, όπως προείπα, έχει πολύ δρόμο για να συμφωνήσει στο εσωτερικό του καταρχήν. Στι ομιλίε με την Προεδρία, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι εμεί να παραλαμβάνουμε τη θέση μα, τη θέση του Κοινοβουλίου. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι είναι υπερβολικά νωρί να συζητήσουμε οτιδήποτε, γιατί δεν ξέρουμε ποια θα είναι η θέση του Συμβουλίου. Πρόεδρο, Πριν ζητήσω από την Κομισιόν τον Ερικ να πει δύο λόγια, ε, ε, θέλ, θέλετε να μιλήσετε μήπως τώρα ή να μιλήσω εγώ. Παρακαλώ. Ειλικρινά δεν ξέρω τι πρέπει να πω σε αυτή τη φάση, γιατί εδώ το θέμα είναι η θέση του, συνοβου... του Κοινοβουλίου και πώς θα διαμορφωθεί σύν το χρόνο. Να μην παρέμβω, αλλά μια που το αναφέρεται να πω ότι η νέα ενδιαμέση κατηγορία, η μετάβαση όπως λέμε, δεν είναι κατηγορία η οποία παίρνει κονδύλια από τις φτωχέ περιοχές για τον εαυτό τη. Δεν παίρνουμε χρήματα από τις φτωχέ περιοχές για να χρηματοδοτήσουμε τη μετάβαση. Αν δείτε την πρόταση της Κομισιόν, θα διαπιστώσετε ότι τα κονδύλια για τι φτωχέ περιοχές και τις περιοχέ. στα νέα κράτη-μέλη αυξάνεται και θα αυξηθεί στο μέλλον σε σύγκριση με την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Και τούτο διότι η χρηματοδότηση προβλέπει μείωση κονδυλίων για την Ευρώπη των 15. Οπότε μην έχετε την εντύπωση σε καμία περίπτωση ότι παίρνουμε λεφτά από τους φτωχού για να τα δώσουμε στις πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης. Όχι, πρόκειται για συνεπή προσπάθεια να ευνοήσουμε τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές στην Ευρώπη. Αυτό. Ευχαριστώ πρόεδρο. Σχόλιο εκτό μικροφώνου. Ιωχήμ, τι και αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα διότι ακόμη και οι πιο πλούσιες λεγόμενες περιοχές υποφέρουν από την κρίση και απλούστατα κανείς δεν το παίρνει είδηση. δεν είπε ότι δεν παίρνουμε λεφτά από τις πιο πλούσιες περιοχές, αλλά δεν έχουμε λύση για όλους. Ούτε επειδή παίρνουμε χρήματα από τις πιο πλούσιες περιοχές, ε, έχουμε χρήματα για τους πάντες. Εν πάση περιπτώσει, για να επανέλθω στον κύριο Κάλφιν, είπαμε ότι θέλαμε από καιρούς καιρών, όχι συνεχώς, ε, να έρχεστε κάθε φορά που συζητάμε το θέμα, να δούμε πώς θα που πηγαίνει, πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Γιατί η Κωνσταντζα μίλησε για μια παραλληλή διαπραγμάτευση. Εμείς ε, μιλούμε για το κανονιστικό πλαίσιο παράλληλα, οπότε επειδή έχουμε διάφορα πράγματα σε αγγείλε, καλό θα είναι να συζητούμε για να μα λέτε πού πηγαίνουμε, πού πηγαίνουν οι διαπραγματεύσει για τον προπολογισμό. γιατί αυτά τα δύο συνδέονται μεταξύ τους. Να συνεχίσουμε λοιπόν να συνεργαζόμαστε. Αντρίου, ε, μάλλον ποιος άλλος θέλει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κάλφιν. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Αν κατάλαβα καλά. Πρώτον, είναι πολύ νωρίς τις διαπραγματεύσεις η διαδικασία επιπλέον δεν είναι σαφής. Δεν έχει αποκρισταλωθεί. Όσον αφορά τη γνώμη μας, βάσει του 3.12 της Συνδίκης της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει τη σύνδεση του με πλειοψηφία των μελών του. Τώρα στην Επιτροπή Προπολογισμών σαφώς πρέπει να συνεργαστούμε με την καθήλυνα αρμόδια Επιτροπή από εδώ και πέρα να έχουμε τακτική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το πώς θα προχωρήσουμε στη σχετική διαδικασία. Και αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την καθήλυνα αρμόδια επιτροπή που θα φροντίσει να γίνει ακουστή η φωνή του Κοινοβουλίου με επιπλέον ε, εκθέσεις, ε, με εκθέσεις της πρωτοβουλίας. Αλλά όπως είπα υπάρχει μεγάλη βεβαιότητα προ την διαδικασία. Θα δούμε πώ θα προχωρήσουμε. Γι' αυτό ευχαριστώ ε, πολύ και χαίρομαι που θα έχουμε συνεργασία τακτική με την Καθήλυνα Αρμόδια Επιτροπή. Πρόεδρο. Ευχαριστώ. Οπότε μπορούμε να κλείσουμε με αυτό. Δεν έχουμε να λάβουμε απόφαση σε αυτή τη φάση. Και άλλο ένα σημείο στην ημερησία διάταξη. Ε, το οποίο δεν έχουμε ποιο τρόπο παρουσιάσει γιατί ο κύριο Φανίστελ Ρόι εξαφανίστηκε. Ε, θα, μιλήσετε, θα μιλήσουμε για την Ελλάδα. Έχετε αξιοδότηση όχι, αλλά επειδή διάβασα την έκθεση, έχω άποψη. Είναι καλή η έκθεση. Αλλά ήδη πέρασαν 4-5 μήνε, τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδιν στην Ελλάδα. Μιλάμε για διαφορετική χώρα σχεδόν. Οπότε ας, σημειώσουμε την ε, έκθεση που λέμε γραπτό και να κλείσουμε. Ναι, δεν χρειάζεται να τη συζητήσουμε δεδομένων των τεράστιων λαών στην Ελλάδα. Σύμφωνα. Δεν χρειάζεται ούτε να εγκρίνουμε τίποτα, Οπότε, αυτοί συνάδελφοι, πολύ ωραία, τίποτα άλλο, στα διάφορα δεν έχουμε οτιδήποτε. Οπότε, 19 και 20 Δεκεμβρίου θα τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.